Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ε, να ξέρετε ότι ε, μεταδίδεται από το διαδίκτυο, του από το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συνεδρίασή μα. Λοιπόν, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Πάμε στο 2 που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης που έγινε στις 15 και 16 Ιουλίου του 2008. Θεωρώ ότι, θα θεωρήσω ότι εγκρίθηκαν εάν δεν υπάρξει αντίρρηση πριν από το πέρας συνεδρίασης. Πάμε στο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου. Θα ήθελα να σας πω ότι ένας κατάλογος με όλη την αλληλογραφία που πήραμε μέχρι σήμερα ε, σας δόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Και όσοι ενδιαφέρεστε για ένα συγκεκριμένο σημείο, σας παρακαλώ να απευθυνθείτε στη γραμματεία της Επιτροπής. Επίσης, να σας πω ότι συμμετείχα σήμερα το πρωί σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας ε, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλίας. Ε, με βάση την πρόσκληση που έστειλε σε μένα και σε όλους τους αντιπροέδρους ε, των ε, επιτροπών ή πρόεδρος. Ακριβώς γιατί θέλουμε ε, το, η διάσταση ισότητα των δύο φύλων να λάβανται υπόψη στις ανταλλαγές απόψεων στα πλαίσια της διετούς έκθεσης που ασχολείται ακριβώς με την συμπερίληψη του θέματος αυτού σε, στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Στην αιτιολογική έκθεση της ε, έκθεσης της κυρίας Ζαμπόρσκα που ήταν η συγγήτρια για την έκθεση αυτή, την ενδιάμεση αυτή έκθεση, συμπεριλαμβάνονται η, συμπεριλαμβάνεται η συμβολή που έστειλε η δική μας Επιτροπή. Στείλαμε ε, τη συμβολή μας μέσω του ερωτηματολογίου που εδόθη σε όλες τις επιτροπές, άρα και στη δικιά μας, και που πήρατε ήδη αντίγραφο. Θα ήθελα απλά και μόνο να σας πω ότι η έκθεση αυτή θα εγκριθεί στην Επιτροπή Γυναικών στις 31 Μαρτίου 2009 και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Απριλίου. Πάμε στο 4, σημείο 4, που έχει να κάνει με τον έλεγχο της υγείας και τη μελλοντική αναθεώρηση της κοινή πολιτικής αλληλείας. Σας θυμίζω ότι το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε καινούρια νομοθεσία ε, ε, σχετικά με το νομικό πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, νομοθεσία που προβλεπόταν για χρονικό διάστημα 10 ετών και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ανάλυση των πρώτων ετών εφαρμογής της νέας πολιτικής για να δούμε ποια ήταν τα ε, δυνατά σημεία και ποια ήταν τα προβλήματα. Για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να χαράξουμε τις κατευθυντήριες γραμμές μιας νέας μεταρρύθμισης το 2012. Οι στόχοι της κοινή αλληλευτικής πολιτικής εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι. Ε, προστασία των πόρων, διατήρηση των ελευτικών πόρων από τη μία, έτσι ώστε να εγγυηθούμε ε, την ε, πραγματική ανάπτυξη των ειδών και την προστασία των οικοτόπων και από την άλλη το μέλλον ενός οικονομικού τομέα που είναι πολύ σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε επίπεδο αγορών όσο και σε επίπεδο εσόδων αλλά και συνθήκων ζωή όλων των εμπλεκομένων στον τομέα. Αλλά και είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά ε, την ίδια τη ζωή των πληθυσμών στι ακτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, είναι προφανέ ότι από το 2000 ε, ε, και εξή είχαμε καλά πράγματα όσον αφορά την επεξεργασία σχεδίων ανάκτηση ή ε, διαχείρισης ορισμένων εμπορικών ειδών, των οποίων τα αποθέματα επαπειλούνται. Ε, σε άλλους τομείς, ε, σε άλλα επίπεδα, όπως για παράδειγμα στο θέμα του ελέγχου. Εδώ πρέπει να δούμε ότι ακόμα ε, έχουν να γίνουν πολλά. Όσον αφορά ορισμένε πτυχέ τη κοινή αλληλευτική πολιτική, εδώ πρέπει να πούμε ότι είχαμε σοβαρέ εξελίξει, όπω για παράδειγμα το ρόλο τη ηχθικολιέργεια για τον εφοδιασμό των αγορών, αλλά και η εξωτερική διάσταση. Όλα αυτά όμω απαιτούν μια ανάλυση σε περισσότερο βάθο για να λάβουμε υπόψη αυτέ τι νέε πραγματικότητε. Η συζήτηση για τον, ε, ε, για τον έλεγχο της υγείας ε, της κοινής ελευθερικής πολιτικής αλλά και για το μέλλον ξεκίνησε από την Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου με, με αφορμή την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Αλίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 όπου συμμετείχε και ο στρατηγός Μοριγιών ως πρόεδρος της Επιτροπής μας. Πρέπει να συνεχίσει λοιπόν αυτό ο προβληματισμός σε ευρύτερη κλίμακα και φέτος θα έχουμε ε, τη δημοσίευση που ήδη ανακοινώθηκε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευση μια πράσινη βίβλου που θα ε, ξεκινήσει μια παρατεταμένη ε, περίοδο δημόσια διαβούλευση το θέμα αυτό. Επειδή είμαστε στο τέλος της θητείας και ε, και, επειδή ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εδώ ε, είναι μικρότερη δραστηριότητα του Κοινοβουλίου, λοιπόν, οι πολιτικοί συντονιστέ τη Επιτροπή μα θέλησαν να εμπλακούν από νωρί σε αυτή την τόσο σημαντική δραστηριότητα και ένα τρόπο είναι και η δημόσια κρόση που έχουμε σήμερα. Έχουμε την ευχαρίστηση λοιπόν να έχουμε και τον Επίτροπο υπεύθυνο για τα αλληλευτικά θέματα και για την Αλία, ο οποίο δέχτηκε να έρθει εδώ και να μα μας ε, βοηθήσει να σχηματίσουμε μία εικόνα για το μέλλον ε, για, το, για, τη μελλοντική πράσινη βίβλο που προβλέπεται να δημοσιευτεί στις 29 Απριλίου. Η, στη συζήτηση επίσης θα, θα έχουμε ε, τη συμβολή εννέα εξεχόντων εμπειρογνωμόνων που, ε, που θα εκπροσωπήσουν τα τρία περιφερειακά συμβουλευτικά συμβούλια και έξι ε, εθνικές διοικήσεις. Καλωσορίζω όλους και θα ήθελα... Ε, να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάζω στο μέτρο που θα παίρνετε το λόγο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Λοιπόν, μετά από την παρουσίαση από τον Επίτροπο Μπόργκ που θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά, θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη ε, της Επιτροπής μας. Οι παρεμβάσεις των υπόλοιπων ε, ομιλητών που θα, θα επιθυμούσαμε να μην ξεπερνούν κάθε μία τα 12 λεπτά θα ομαδοποιηθούν σε, τρία, σε τρεις ενότητες. Μετά από κάθε ενότητα θα αφήσουμε το, το χρόνο για τη συζήτηση. Ο Επίτροπος Μπόργκ μας είπε ότι μετά ε, την ε, παρέμβασή του και την ανταλλαγή των απόψεων ε, που θα ακολουθήσει είναι υποχρεωμένος να φύγει. Αλλά θα έχουμε εκπροσώπους Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ οι οποίοι θα είναι παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίασης για να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής μας ή για να τοποθετηθούν στις διάφορες παρεμβάσεις. Να δώσω λοιπόν τον λόγο πρώτα απ' όλα στον Επίτροπο Μποργ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω όλους που μου δίνετε την ευκαιρία που οργανώσατε τη σημερινή συζήτηση για να συζητήσουμε το μέλλον της κοινή πολιτικής αλληλείας. Οι παλιότερες συζητήσεις που κάναμε εμπλούτησαν την γενικότερη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση και σίγουρα σήμερα θα γίνει το ίδιο. Η κοινή δουλειά που κάναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια για να βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα και να καταλήξουμε σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον υγιεινό για να μπορέσουμε να κάνουμε την ε, αλία μας βιώσιμη άρχισε να αποδίδει καρπούς και πραγματικά είναι ε, αποτέλεσμα της ε, αφοσίωση την οποία δείξατε κι εσείς παρόλο όμως που έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερα και υπάρχουν πολλά ειδικά θέματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Γι' αυτό το Συμβούλιο πρόσφατα ενέκρινε την, τον κανονισμό IUU και γι' αυτό η Κομισιόν υπέβαλε και μια πρόταση για να αλλάξει, να αναθεωρήσει την πολιτική ελέγχων της κοινή πολιτικής αλληλείας για να γίνει η διαχείριση πιο αποτελεσματική και να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες. Αργότερα θα υποβάλουμε μια πρόταση για να μεταρρυθμίσουμε ρυθμίσουμε την κοινή οργάνωση αγοράς. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σημαντικές και μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης και στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων. Όμως η πετρελαϊκή κρίση και η, οικονομική κρίση στην, την οποία διατρέχουμε έδειξαν πόσο δύσκολο είναι να έχει κανείς μια σταθερή οικονομική βάση για την για τον αλλιευτικό κλάδο και επίπεδα κερδών που θα μπορούσαν να κάνουν βιώσιμη την δραστηριότητα αυτή. Διαρθρωτικές αλλαγές λοιπόν είναι αναπόφευκτες μετά το τέλος της κρίσης και ο κλάδος θέλουμε να, γιατί ο κλάδος θέλουμε να γίνει βιώσιμος μακροπρόθεσμα. Πρέπει να Πρώτα βέβαια να βγούμε από την κρίση όταν η αλληλεία μειώνεται συνεχώς ή μάλλον οι αλληλευτικοί πόροι μειώνονται συνεχώς και ούτω τα κέρδη πέφτουν και πολλοί αλληλείς και ολόκληρες παράκτιες κοινότητες πληθυσμιακές αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Το περιβάλλον επίσης πρέπει να μας σταματήσουμε την υπεραλίευση των πόρων μας, την απόρριψη ηχθείων και πρέπει να επανέλθει η παραγωγικότητα στους ωκεανούς και στις θάλασσές μας. Δεν ναι, είναι μόνο οικολογικοί οι λόγοι που μας επιβάλλουν κάτι τέτοιο, είναι και ηθικοί οι λόγοι και τα μακροπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα του αλλιευτικού τομέα το απαιτούν αυτό. Επίσης η εμπορία των αλλιευτικών προϊόντων πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Χρειαζόμαστε επίση πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην, ε, ε, στο εμπόριο και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Ένα τέτοιο εργα, εργαλείο που έχουμε εδώ είναι το λεγόμενο eco-labeling και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μελετούν μια πρόταση της Κομισιόν αυτή τη στιγμή για την οικολογική αυτή σήμανση και ένα σύστημα Community Eco-Label Award ε, θεωρήσαμε ότι σε αυτό το σύστημα πρέπει να ενταχθούν και αλληλευτικά προϊόντα και βεβαίως ε, ελπίζουμε να περάσει η πρότασή μας αν όμως δεν περάσει θα προτείνουμε ένα ειδικό σύστημα για οικολογική σήμανση ειδικά για τον τομέα της όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εξαρτώνται βεβαίως από το πόσο θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί η η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιζήσει χωρίς κοινή πολιτική αλληλείας. Το θέμα δεν είναι να επανεθνικοποιηθεί η πολιτική αυτή όπως λένε ορισμένοι. Δεν θέλουν, γιατί η πολιτική αυτή, η αλληλεία βασίζεται σε πόρους οι οποίοι είναι κοινοί. Εκείνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να πλουστεύσουμε και να μεταρρυθμίσουμε εκ βάθρων την πολιτική αλληλείας πρέπει να φτιάξουμε μια πολιτική κατάλληλη για τον 21ο αιώνα. Μια πολιτική που θα βοηθήσει τον κλάδο να ε, κάνει κέρδη, να μπορεί να αυτονομηθεί οικονομικά και να παράγει υγιεινά και ασφαλή ε, τρόφιμα στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Μια πολιτική που να προστατεύει το περιβάλλον και να είναι βιώσιμη. Να, μια πολιτική που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ανάπτυξη των που θα βοηθήσει τον κλάδο να αισθάνεται ασφαλής και που θα είναι αποτελεσματική απλή στην εφαρμογή της και θεμητή και, και για τον, ε, τους αλείς και για τους πολίτες της Ένωσης. Ξεκινώντας λοιπόν τη διαδικασία μεταρρύθμισης νωρίς και προσπαθώντας να την περάσουμε σε ε, μια όσο πιο ευρεία βάση γίνεται και ζητούμε τολμηρές λύσεις για να χαράξουμε ένα δρόμο που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε την αλία μας μακροπρόθεσμα. Το, η πράσινη βίβλος που θα εκδοθεί πραγματικά και που θα παρουσιαστεί αναλύει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή παρουσιάζει το όραμα προς το μέλλον και αυτή τη στιγμή είμαστε τελείως ανοιχτοί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε και άλλα στοιχεία της πολιτικής που είναι εδρεωμένα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε βασικά προβλήματα Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιους βασικούς στόχους όλοι μας. Πρώτος στόχος, μια πολιτική αποτελεσματική, απλή και η εύκολη στη διαχείρισή της. Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται σε ένα επίπεδο κοντά στον κόσμο που επηρεάζεται. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να αναθέσουμε περισσότερη ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων στα κράτη-μέλη, στην Κομισιόν και υπό συγκεκριμένου όρους στον ίδιο το κλάδο. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας υποστηρίξει στο στόχο αυτό και θα συνεργαστεί με την Κομισιόν για να φτιάξουμε μια τέτοια κοινή πολιτική αλίας. Δεύτερος στόχος, ο κλάδος πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά και ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε κάτι τέτοιο είναι να δώσουμε στους αλείς περισσότερη ευθύνη. Έγιναν πρόοδοι στον τομέα από το 2002 ε, και δόθε ωστόσο η βασική φιλοσοφία της πολιτικής αλίας παραμένει εκ των άνω προς τα κάτω οι ενδιαφερόμενοι αυτή τη στιγμή δεν αισθάνονται ότι συμμετέχουν αρκετά για να χαράξουν πολιτική και Πιστεύουμε βεβαίως ότι ο καινούριο κανονισμός IUU και οι πρωτοβουλίες που πήραμε για τον έλεγχο θα με αλλάξουν κάπως τη φιλοσοφία ή την προσέγγιση μας αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη ενεργό συμμετοχή του κλάδου των αλλιέων αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας υπάρχουν παραδείγματα βεβαίως όπου ο ίδιος ο τομέας ανέλαβε την εφαρμογή της πολιτικής αλλίας και τα παραδείγματα αυτά είναι ενθαρρυντικά. Υπάρχουν οργανώσεις παραγωγών που επιτυχώς ανέλαβαν τη διαχείριση ποσοστώσεων. Αυτή η αυτοδιαχείριση αν θέλετε του κλάδου θα πρέπει να πάει πιο πέρα να, γι, να θεσμοθετηθεί σχεδόν και Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε και τον κλάδο να υιοθετήσει ουσιαστικά την πολιτική και να θα τον υποκινήσει να αναπτύξει τις δικές του λύσεις στα προβλήματα σε, ένα μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο. Επίσης πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια είναι μία από τις ε, μεγάλες επιτυχίες της μεταρρύθμισης του 2002 και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ούτως ώστε να υπάρχει διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Και έρχομαι τώρα στον τρίτο ε, στόχο. Ε, περιφερειοποίηση τρόπον την της ε, κοινή πολιτικής αλίας. Ε, δια, η, χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική όπου θα βασιζόμαστε στις ίδιες αρχές για οικονομική, οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα μόνο αν πιστεύουμε όλες τις ίδιες αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο θα, μπορούσαμε να θα μπορούμε να δουλέψουμε όλοι με ίσους όρους συγχρόνως όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι θάλασσές μας και οι αλίες μας είναι τόσο πλούσιες ακριβώς επειδή είναι τόσο διαφορετικές δεν μπορούμε να ε, πέρα από τις γενικές αρχές δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε όλα τα ίδια πράγματα, τις ίδιες λύσεις. Και η, αυτή τη στιγμή που εφαρμόζουμε ουσιαστικά ένα κεντρικό micromanagement ε, δημιουργούμε προβλήματα, αντί να τα λύνουμε. Το να επέμβουμε λοιπόν, να περδένουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα θέματα είναι λάθος και δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει και με τη μελλοντική εφαρμογή της συναπόφα, διαδικασίας συναπόφασης. Γι' αυτό υπάρχουν σοβαροί θεσμικοί λόγοι και ε, η κοινή λογική λέει ότι πρέπει να βρούμε ε, λύσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εφαρμόζουμε αποφα... να παίρνουμε αποφάσεις στο σωστό επίπεδο και να τις εφαρμόζουμε στο σωστό επίπεδο και αυτό σημαίνει κατάτμιση αν θέλετε της θάλασσας μας σε περιφέρειες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη δουλειά αυτή μέσα σε συνεργασία με τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια στη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Επίσης πολλά από τα θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα θα περάσουν στο ε, προοδευτικά θα περάσουν στη λεγόμενη ναυτιλιακή πολιτική ε, και αυτό αμέσως θα ξεχωρίσει τα πράγματα και ένα παράδειγμα για το τι μπορούμε να κάνουμε είναι η, μια οδηγία που εγκρίθηκε ε, πρόσφατα στο πυλώνα του περιβάλλοντος ε, της στρατηγικής της θάλασσας Marine Strategy Directive η οποία ουσιαστικά η οποία θέτει ε, περιφερειακούς ποιοτικούς στόχους που βεβαίω πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη γενική πολιτική αλληλεία. Τώρα, ο τέταρτο και τελικός στόχο ε, της ε, πολιτικής σχετίζεται με τον εξωτερική διάστασή τη. γιατί βεβαίω ε, οι στόχοι πέρα από τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και τα παγκόσμια ύδατα και υπάρχουν και ανηλυμένες διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορέσουμε ε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή μια βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας καλή διακυβέρνηση των θαλασσών και των ωκεανών θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να βρούμε τρόπους να ε, είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στη ε, καταπολέμηση μη θεμητών δραστηριοτήτων και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος ε, είπαμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή και τη χρήση των διμερών συμφωνιών για να μπορέσουμε να ε, προωθήσουμε τις επενδύσεις της Ένωσης σε τρίτες χώρες και να ενισχύσουμε το δυναμικό μας στις αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορούμε τελικά να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα ε, τους φυσικούς πόρους και θα πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς μεταξύ των περιφερειακών και διμερών προσεγγίσεων της πολιτικής μας. Όλα αυτά που ανέφερα κυρίες και κύριοι είναι κάποια από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε ε, πριν να αποφασίσουμε για τη μεταρρύθμιση κοινή πολιτικής αλίας. Η πράσινη βίβλωση η οποία θα δημοσιευθεί νομίζω ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από όλους σαν βάση για μελλοντικές πολιτικές συζητήσεις θα ελπίζω ότι θα δώσει κίνητρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, τους πολίτες, προσώπους τους ε, οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν για να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε μια καλή ε, κοινή πολιτική αηλία στο μέλλον. Έχουμε μια σημαντική ευκαιρία μπροστά μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σε διαρκή βάση και θετικά τα πράγματα. Και πριν να κλείσω την παρέμβασή μου θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για την, τον, την πρόταση που κάναμε για, την, για τους ελέγχους στην πρότασή μας περιλαμβάνεται ο όρος αλληλεία αναψυχής. Σε κάποια κράτη-μέλη πρότασής μας παρεξηγήθηκαν και ξεσηκώθηκαν οι εραστέχνες ψαράδες οι οποίοι έχουν σαν χόμπι την αλία και φαντάστηκαν ότι η Κομισιόν θα αρχίσει να τους κυνηγά. Προφανώς θα ήταν τρελό να προτείνουμε κάτι τέτοιο και που δεν είναι λόγο θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο γελίο σύστημα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω λοιπόν μια και καλή ότι ο ερασιτέχνης ψαράς που πιάνει μερικά κιλά ψάρι κάθε λίγο και λιγάκι και τα χρησιμοποιεί για το βραδινό του τηγάνι δεν πρόκειται να ε, καλύβεται από τον κανονισμό μας ακόμη και αν ψαρεύει μπακαλιάρο ε, υπάρχουν όμως στοιχεία και νούμερα τα οποία μας δείχνουν ότι αρισμένες μορφές αλίας αναψυχής ε, έχουν επιπτώσεις και μάλιστα επικίνδυνες επιπτώσεις σε κάποιους αλλιευτικούς πόρους. Γι' αυτό δεν μπορούμε από τη μια στον επαγγελματία ψαρά να επιβάλλουμε περιορισμούς και στον εραστέχνη ψαρά να αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο. Θα πρέπει και ο εραστέχνης ψαράς να συμβαίνει συμβάλλει. Με αυτή την έννοια λοιπόν αναφέρουμε τον όρο αυτό στην πρότασή μας και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, με από ανυπομονησία περιμένουμε να συνεργαστούμε για τα θέματα αυτά μαζί σας για το όλο θέμα των ελέγχων και του σχετικού κανονισμού για την όλη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής αλίας. Εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι εμείς στην Κομισιόν μπορούμε πάντα να βασιστούμε στο Κοινοβούλιο και τώρα είμαι στη διάθεσή σας κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε να απαντήσω ερωτήσεις αν και εφόσον υπάρχουν. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Αυτή τη στιγμή έχω 7 στον κατάλογο μου. 7 συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν και θέλουν να σα υποβάλουν ερωτήσει. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ μία πρώτη ερώτηση, επί τη διαδικασία, ε, Επίτροπε. Η πρώτη μου ερώτηση, ή μάλλον η ερώτησή μου είναι η εξή. Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η περίοδος διαβούλευσης, ε, μόλις δημοσιευθεί η πράσινη βίβλος, ένα χρόνο, λίγους μήνες, γιατί εμείς θα διαρκεσει η περιοδο διαβουλευση ε μολις δημοσιευθει η πρασινη βιβλο ενα χρονο λίγου μήνε, γιατι εμεις θα θελαμε να ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στην κυρία Φράγκα, ναι. εξ ονόματος του ΕΛ. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε σήμερα να μας παρουσιάσει τις πρώτες του ιδέες για την μεταρρύθμιση της ε, κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ε, Επίτροπε δεν θέλω να μακρηγορήσω. Γιατί, τι να σας πω, κάθε θέμα που θίξατε χρειάζεται μια συζήτηση από μόνο του. Θα ήθελα πάντως να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Εντάξει, πολλές φορές ε, ε, απευθύνουμε κριτικές. Αλλά ε, σας ευχαριστούμε γιατί πραγματικά τολμήσατε να ξεκινήσετε με σοβαρότητα μια μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση του μοντέλου διαχείρισης. Ε, θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση του 2002 ήταν μήνυ μεταρρύθμιση. Γιατί το βασικό πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην κοινή πολιτική τα τελευταία χρόνια προέρχεται από το σύστημα των ΤΑΚ και ποσοστώσεων ε, και από την αρχή τη σχετική σταθερότητα. Δεν σα το λέω εγώ. Όλε οι προκαταρκτικέ μελέτε ε, ε, που αναθέσατε εσεί σε Ισπανού αλλά και σε μία σειρά άλλου εμπειρογνώμονε από όλα τα πεδία, όλε λοιπόν οι μελέτε δείχνουν αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ακριβώ το μοντέλο διαχείριση το οποίο είναι παροχημένο. Και όλα τα προβλήματα, ακόμα και τη ε, υπεραλίευση, ακριβώ προέρχονται από το υφιστάμενο μοντέλο διαχείριση. Λοιπόν, πριν από τη μεταρρύθμιση 2002, ήδη στο Κοινοβούλιο είχαμε ε, ε, αναφέρει πολλέ ιδέε. Να μιλήσουμε για δικαιώματα αλληλεία, ε, να μιλήσουμε για τη διαφορά ανάμεσα στη βιομηχανική αλληλεία και στη βιοτεχνική κτλ. Πάντω αυτό είναι ο μοναδικό δρόμο που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με σοβαρότητα για να δούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η αλληλεία. Και αναφέρω και το πρόβλημα τη υπεραλίευση. Διότι είναι σαφέ ότι η αρχή τη σχετική οικονομικής ε, σταθερότητας ε, ε, προσεγγίζει το θέμα μόνο από την άποψη της αγοράς. Και πραγματικά δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά και κοιτάξτε γίνονται μια σειρά από συζητήσεις στα κρατημέλη, ακούγονται και οι απόψεις του κλάδου, άρα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Χωρίς βεβαίως να, να τιμωρήσουμε υπερβολικά τους μεν τους δε, πρέπει όμως να φέρουμε μια λογική. Χωρίς να γίνει αυτό τα υπόλοιπα δεν έχουν νόημα. Τώρα, τούτου λεχθέντος, ε, και ακριβώ ε, τονίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σα πω ότι ε, τόσο όσον αφορά τι μελέτε τι οποίε αναθέσατε στου εμπειρογνώμονε, αλλά και από τι πρώτε σα απόψει, εκεί που νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα είναι ε, η εξωτερική πολιτική. Και γιατί σα το λέω, Γιατί πιστεύω ότι η ανάλυση δεν, δεν χαρακτηρίζεται από τον ρεαλισμό. Ε, αναφέρονται διάφορε αντιλήψει που υπάρχουν, αλλά αυτό έχουν να κάνουν με τι αντιλήψει μια μερίδα των πολιτών, που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι οι πλέον εμπλεκόμενοι στο τομέα. Αλλά εμένα με απασχολεί κυρίω το θέμα των διμερών αλληλευτικών συμφωνιών. Γιατί, λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα οποία διάβασα από τα λίγα έγγραφα ε, που διαθέτουμε για το θέμα, εσεί όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και τι διμερεί ε, συμφωνίε, θέτεται προτεραιότητα σε μια εξωτερική πολιτική που να ε, ευνοεί τις επενδύσεις σε τρίτες χώρες. Επίτροπε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι η πολιτική. Αν μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική. Εγώ θα ήθελα να μάθω τι πιστεύετε πραγματικά όσον αφορά το μέλλον των διμερών συμφωνιών αλίας ή των ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Πιστεύετε ότι πρέπει να τη συνεχίσουμε ή από ό,τι φαίνεται ε, και όπως διαφαίνεται λαμβάνοντα υπόψη και ορισμένου στόχου που θέτετε εσεί σε αυτά τα πρώτα έγγραφα, φαίνεται ότι θέλετε να καταργηθούν αυτέ οι συμφωνίε. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Φράγκα. Κυρία Άτγουλ, έχει το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Τρία θέματα θέλω να σχολιάσω. Πρώτον, την αυτά που την ανακουφίση με την οποία θα χαιρετήσουν οι ερασιτέχνες ψαράδες αυτά που είπατε σχετικώς. Διότι η πρόταση έτσι όπως έχει διατυπωθεί στο σημείο 47 μπορεί πράγματι να παρερμηνευτεί. Ο κ. Ρωμέβα ήδη έχει προτείνει τροπολογίες για να αποσαφινιστούν τα πράγματα και ελπίζω η Κομισιόν να δεχτεί να ακούσει τουλάχιστον τα σχόλια του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δεύτερο, οι οικομάρκες ή οικοετικοτοποίηση. Ξέρω ότι υπάρχει η οριζόντια οδηγία που συζητάται αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον πρέπει και η αλληλεία να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον σύμφωνα με μια από τις κοινοβουλευτικές μας επιτροπές. Εγώ προσωπικά και το λέω, το τονίζω ότι το λέω προσωπικά είναι ότι είναι τόσο πολύπλοκη η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος οικομαρκών στην αλληλεία ώστε θα ήθελα λίγα περισσότερα σχόλιά σας. Και τρίτον, συμφωνώ ότι αν υπάρξει μεταρρύθμιση και υπάρξουν ουδέτερες ζώνες τότε πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει παρόλα αυτά κάποια ισορροπία γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αλλιευτικές κοινότητες που εδώ και πολλές γενιές εξαρτώνται από την αλία, από την αλλίευση ορισμένης ποσότητας ψαριών και αν δεν προσεχθούν σύμφωνα με το σχέδιο αυτό δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν οι κοινότητες αυτές και μάλιστα θα επηρεαστεί ολόκληρη η οικονομία της περιφέρειάς τους γενικότερα. Ελπίζω όμως η Κομισιόν να το προσέξει και να μην βλάψει ιδιαίτερα την μικρών διαστάσεων τοπική αλληλεία, αλλά να δει το πρόβλημα γενικότερα. Θα ήθελα λοιπόν και από αυτού ορισμένα περισσότερα σχόλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Άτγουλ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κασάκα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον Επίτροπο για την εισήγησή του Δύο κύρια στοιχεία έχω δει ότι έλειπαν από την εισήγηση όμως αυτήν και θα ήθελα να μου πει τι φρονεί για αυτά. Πρώτον, κατά, σε τι βαθμό θα λάβει υπόψη του την κατάσταση που επικρατεί σε απομακρυσμένες περιοχές και δεύτερον, πώς σκοπεύει να συνδυάσει τα οικοσυστήματα με την αλληλεία γενικότερα. Τώρα για την ερασιτεχνική αλληλεία νομίζω ότι το σύστημα που προτείνεται μπορεί να μην το βλέπουμε με, τον ίδιο τρόπο εμείς και η Κομισιόν. Α, έχει δίκιο βασικά η Επιτροπή ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τελείως τα πλαίσια της ΚΑΟΠ την ερασιτεχνική αλή, αλλά ιδιαίτερα δεδομένου του ότι χάνουμε μεγάλες ποσότητες αλληλευμάτων. Ευχαριστώ τον κύριο Κασάκα. Να δώσω το λόγο τώρα ε, στον κύριο Χάστον. Ε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ επίτροπε που ήρθατε εδώ και η οποία με χαροποιεί κάθε φορά αυτή τη φορά όμως ναι. δεν χάρηκα με όλα αυτά που είπατε ε, τονίσατε ορισμένα πράγματα για την μεταρρύθμιση της μελλοντική κοινή πολιτική αλληλείας και είπατε ότι θα πρέπει να γίνει εκβάθρονη αλλαγή αυτή. Αλλά εγώ δεν ε, νομίζω ότι ε, ε, αυτό είναι, νομίζω όμως ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν τα ακούει κανείς έτσι. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να, λύσει, να επιβιώσει χωρίς κοινή πολιτική αλληλείας. Εγώ θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κάλλιστα να ζήσει δίχως την κοινή αυτή πολιτική. Η κοινή πολιτική αλληλείας ε, συμφωνήθηκε κάποτε, συμφωνήθηκαν και κάποιοι στόχοι οι οποίοι όμως δεν ποτέ. Και το μόνο που έγινε είναι ότι σε ορισμένε περιοχές των υδάτων μας δεν μπορούμε να αλλιεύσουμε. Εγώ δεν ξέρω τώρα τι θα πει μεταρρύθμιση. Θα αναθεωρήσουμε ε, αυτά που λέμε στην τωρινή κοινή πολιτική αλληλείας που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτή και ίση πρόσβαση σε όλες τις περιοχές για όλους αν ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε ανησυχώ διπλά ένας άλλος λόγος που Εμείς που δουλεύουμε στον κλάδο ανησυχούμε είναι ότι πρώτον εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα πρέπει να αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τους ολιευτικούς πόρους από τους οποίους ζούμε. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να σεβόμαστε τους αλληλευτικούς πόρους και η ίση και ανοιχτή πρόσβαση όλων παντού νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο θα παραμείνει θα πρέπει να παραμείνει είναι λοιπόν μεγάλη απειλή το να ε, λέγεται ότι όλα αυτά θα αλλάξουν θέλω να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν τι λέτε διότι αν δεν εννοείται πραγματική εκβάθρον μεταρρύθμιση η μεταρρύθμιση αυτή προτείνεται δεν είναι ε, ιδιαίτερα μεγάλη και σημαντική λέτε εδώ τώρα μεγαλύτερη ε, περισσότερες εξουσίες στα κράτη-μέλη είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο εγώ νομίζω ότι οι φυστάμενοι κανόνες και κανονισμοί και ε, η φυστάμενη συνθήκη αποκλείει την ανάθεση ευθυνών και εξουσιών στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν η συνθήκη της Λισαβόνας θα αλλάξει τα πράγματα. Επίσης, δεν ξέρω τι εννοείται ε, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των αρχών που ήδη υπάρχουν των περιφερειακών συμβουλίων κλπ. κλπ. Δηλαδή θα παίρνουν όλες τις αποφάσεις οι αρχές αυτές. Ευχαριστώ κύριε Χάστον. Να δώσω το λόγο στον κύριο Στίβενσον, να σας θυμίζω ότι έχουμε 8 ομιλητές που θέλουν ακόμα να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να είστε λίγο πιο σύντομοι. Κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο για αυτά που μας είπε για την ερασιτεχνική αλληλεία. Το είπαν και άλλοι, είναι πολύ καλό νέο αυτό που μας ανέφερε Εξάλλου στην πρόσφατη δημοσίευση της Επιτροπής που αναφέρεται στους Καρχαρίες ε, τα είχε ήδη αναφέρει η Επιτροπή αυτά τα καθησυχαστικά στοιχεία. Αφού όμως μιλάμε για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απλοποίηση των συστημάτων, ίσως να χρειάζεται, όπως είπατε και εσείς, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα της λιγότερης κεντρικής διαχείρισης ή μικροδιαχείρισης και όπως είπε και ο κύριος Χάτσον αν θα μπορούσε να γίνει αυτό μέσω της μεταφοράς περισσότερων δικαιοδοσιών στα περιφερειακά συμβούλια αυτό θα ήταν όντως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος και πραγματική πρόοδος. Αλλά βέβαια την μεταρρύθμιση αυτή πρέπει πάντοτε να τη βασίζουμε σε κάποια γενικότερη πολιτική και μέχρι τώρα η πολιτική αυτή στην οποία βασίζεται η πρόταση έχει αποτύχει γιατί στοχεύει μόνο στη διατήρηση των αλλιευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θέσεων εργασίας στην σχετική βιομηχανία αλλά δεν τα κατάφερε ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Βλέπετε πόσα είδη κινδυνεύουν από εξαφάνιση και πόσες χιλιάδες θέσεων εργασίας έχουν απολεσθεί. 60% του αλλιευτικού στόλου του Ηνωμένου Βασιλείου ε, έχουν καταστραφεί τα τελευταία χρόνια. Και η μόνη μέθοδος που προτείνουμε είναι να μειώσουμε τα αλλιεύματα. Και βέβαια κατηγορούμε πάντοτε τους αλληλείς, αλλά δεν εξετάσαμε ποτέ μήπως δεν έφταιγε η ίδια η ΚΑΛΠ. Εκείνη νομίζω εγώ ότι φταίει για την καταστροφή αυτή. Η μεταρρύθμιση λοιπόν σίγουρα χρειάζεται και είναι πια καιρός να εφαρμοστεί, αλλά το πρόβλημα είναι με ποιο σύστημα διαχείρισης θα εφαρμοστεί. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα ελέγχου, φορολογικά, ποσοστώσεις και άλλα. Δεν θα μπορούσαμε καταρχήν να καταργήσουμε τις ποσοστώσεις και να γίνει ένας πιο συγκεντρωτικός έλεγχος των προσπαθειών περιορισμού των αλλιευμάτων ώστε να μην ζημιώνουν οι ίδιοι οι αλληλείς ενώ φταίει το διαχειριστικό μας σύστημα. Αυτή η πολιτική ε, προσπάθειας μείωσης των αλλιευμάτων και πώληση όλων των αλλιευμένων ψαριών χωρίς να πετιούνται στη θάλασσα ορισμένα θα ήταν κάποια λύση. Και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους μικροαλληλεί σε τοπικές αλληλευτικές κοινότητες, απομακρυσμένες αλληλευτικές κοινότητες. Τέλος, εισάγουμε 60 με 70% των ψαριών που καταναλώνουμε στην Ένωση, αλλά δένουμε τα χέρια των ηχθειοκαλλιεργητών μας με εκατοντάδες κανονισμών από πάρα πολλές γενικές διευθύνσεις, ΣΑΝΚΟ, ΕΝΒΙ, ΜΑΡΙ. Ίσως αυτή τη μεταρρύθμιση θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και ένα καλύτερο σύστημα ελέγχου, δηλαδή τα επόμενα πέντε χρόνια μετά τις εκλογές, να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα ελέγχων των παραγωγών εκτός ένωσης, όχι μόνο των δικών μας, τότε μόνο θα υπάρχει η συμμεταχείριση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Λοιπόν, σα ξαναθυμίζω ότι πρέπει να είστε λίγο πιο σύντομο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Άλιστερ. Σα ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, στην, στα πολλά θέματα που θίξατε, πρέπει να σα πω ότι απογοητεύτηκα γιατί δεν άκουσα καμία αναφορά σε σχέση με το σκάνδαλο των απορρίψεων. Γιατί αν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αμάβρωσε την εικόνα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, και ε, Πραγματικά, αν είναι κάτι, ε, είναι αυτό το θέμα των απορρίψεων. Ορισμένοι από εμά πέρσι επισκεφθήκαμε την Νορβηγία. Και νομίζω τώρα εντάξει, μιλώ σε προσωπική βάση, αλλά νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι εντυπωσιάστηκαν από ε, το πώς, από τις δραστηριότητες της βιομηχανίας εκεί, όπου ο κανόνας είναι ακριβώς το αντίθετο από τη δική μας την πολιτική από εδώ που ήρθα εγώ στην Επιτροπή πριν από πέντε χρόνια μιλάμε για το ίδιο θέμα και εξακολουθούμε να μιλάμε. Εξακολουθούμε να συζητάμε. Εξακολουθούμε να μιλάμε για βελτίωση των πραγμάτων. Και όμω είναι ε, ε, ένα από τα κατάφορα παραδείγματα ε, που δείχνει τα προβλήματα, τα διαρκή προβλήματα στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Μιλήσατε για βιώσιμη αλληλεία. Αλλά όπω είπε ο κύριο Στίβενσον, η κοινή αλληλευτική πολιτική στην ουσία είναι μια πολιτική που έχει αποτύχει. Αν πάρω τη δική μου την ε, περιοχή, να οποία τη γνωρίζω, και δούμε ε, τι γίνεται με το στόλο. Και δούμε τι γίνεται με τα, με λευκά ψάρια. Ε, να δούμε τι έγινε με το σύστημα ανάκτησης του βακαλάου, τους περιορισμούς κτλ. όλα τα προγράμματα είχαν ως στόχο την ανάκτηση. Σήμερα με όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε πετύχει την ανάκτηση των αποθεμάτων. Ε, με αυτό δεν είναι ένδειξη αποτυχημένης πολιτικής. Και καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση όπου αντί για 40 ε, πλοία ε, να ε, μιλάμε για 6. Όταν μιλάμε δηλαδή για πολλά πλοία τα οποία αλλιεύουν λίγα ψάρια, τότε τι λέμε. Τι, λέμε, τι να πω εγώ στους ψηφοφόρους μου, να πω να εγκαταλείψουν την αλία των λευκών ψαριών, να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό είναι ο βασικός στόχος της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Γιατί ε, από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει. Επίσης, να σας πω και να υποστηρίξω το εξής. Εάν θέλουμε η μεταρρύθμιση να έχει νόημα, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να φύγει είναι τα τάκ και οι ποσοστώσεις. Έχουμε αυτή την διαχείριση εκ των άνω προς τα κάτω και τα πράγματα ε, οδηγούν σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε στην πράξη. Και στη συνέχεια έχουμε περαιτέρω διαχείριση της αλλιευτικής ικανότητας, ημέρες στη θάλασσα κτλ. Και τελικά το σύστημα αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Απευθύνω έκκληση λοιπόν. Τα, τα και οι ποσοστώσεις πρέπει να φύγουν. Και είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδείξει ανοιχτή στάση προς το θέμα αυτό και θα ε, δεχθεί την άποψη αυτή. Ευχαριστώ. Επιμένω. Πρέπει να είστε πιο σύντομοι. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ρωμέβα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη που έχει να κάνει με την παρέμβαση του Επίτροπου Μπόρκ και σε σχέση με τη μείωση της ικανότητας, ελευτικής ικανότητας των στόλων. Το αναφέρατε εν παρόδο, αλλά εγώ θα θέλω, θα να σας ρωτήσω το εξή. Μπορείτε να μας πείτε προς ποια κατεύθυνση σκέφτεστε ότι πρέπει να κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Ε, και επίσης, τι γίνεται με τα κοινωνικο-οικονομικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε ε, να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα προβλήματα που ε, πλήττουν ε, ορισμένους. Και, έτσι να, και να πω και το εξή, όσον αφορά την έκθεση ελέγχου ε, που, είναι, που κάνουμε εμεί σε αυτή την επιτροπή. Πράγματι, η αλία για ψυχολογικού λόγου θα αποτελέσει κεντρικό ε, θέμα στη ζήτηση. Το συζητάμε το θέμα με διάφορε ε, ε αντιπροσωπείε για να βρούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που είπε ο κ. Μόργκ. Ε, πραγματικά δεν θα πρέπει να υπάρχουν αμφιλεγόμενα στοιχεία και, να καταλήξουμε, και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ικανοποιητικά κείμενα. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να ε, μα απασχολήσουν και να είναι το επίκεντρο του κειμένου. Σας ευχαριστώ όχι μόνο για την επικοδομητική στάση ε, τη Επιτροπή, αλλά και του άλλου συναδέλφους ε, και τι οργανώσει. Όλοι μα βοηθούν για να επιταχύνουμε τις εργασίες μας για την έκθεση αυτή. Γιατί όπως ξέρετε, ε, εδώ τα πράγματα ε, και ο χρόνος πιέζουν περισσότερο σε παιδοκοινοβουλίο έναντι του χρόνου που έχει διαθέσει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην κυρία Ντόιλ. I'd like to join the thanks to Commissioner Borg. Um, is ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόργκ που βρίσκεται εδώ και πραγματικά είναι παραδειγματικός ως Επίτροπος ε, στη γενναιοδορία του χρόνου που μας διαθέτει. Ε, θα ήθελα τώρα να πω ότι σημείωσα και το πιστεύω αυτό που λέτε ότι είστε ανοιχτοί και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην μπορείτε να αναθεωρήσετε ενδεχομένω σχέση με αυτά που αποφασίστηκαν παλιά. Ωραία, αν Υπονοείται και είναι γεγονός ότι βεβαίως αν φτιάχναμε τώρα την κοινή πολιτική αλληλείας δεν θα κάναμε αυτό που κάναμε δεκαετία του 70 ε, άρα δεν θα υπήρχαν και τάξ και κουότας και ποσοστώσεις πραγματικά η επουδενή λόγο ο κλάδος μπορεί να σας να δεχθεί ε, ε, την ε, επιχειρηματολογία η οποία οδήγησε στα maximum επιτρεπόμενα αλλιεύματα και στις ποσοστώσεις της δεκαετίας του 70. Ο κλάδος είναι υπεύθυνος, δεν θέλει να φτωχύνουν οι αλλιευτικοί πόροι που δεν είναι λόγο. Ρωτώ λοιπόν, η βασική ιδέα των τάξ και των ποσοστώσεων της παλιάς κοινής πολιτικής αλληλείας Αμφισβητείτε την πετάμε στα σκουπίδια να κάνουμε κάτι καινούριο διότι αν δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν κάνουμε τίποτα η βασική αρχή αυτή λοιπόν που διείπε την παλιά κοινή πολιτική αλληλείας και η οποία θεωρείται άδικη αυτή τη στιγμή καταργείται αυτή είναι η κατάσταση Επίτροπε και αυτό είναι το βασικό θέμα κύριε Επίτροπε. Τώρα για την... ήμουν εισηγήτρια για την Επιτροπή αυτή για το θέμα των απορρίψεων και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ε, κοινή αλλοευτικής πολιτικής εδώ είναι πραγματικά οι χιλιάδες τόνοι που απορρίπτονται θεωρούνται παραλίευμα οι ηχθείς αυτοί και πρέπει να πεταχτούν διότι αλλιώς είναι παράνομος ο αλλιέας που τα διατηρεί. Οι απορρίψεις λοιπόν είναι σκάνδαλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ε, αυτό ισχύουν οι κανόνες για τις απορρίψεις, το κατά πόσο υπάρχει θέμα μεγέθους και τα Τέλος πάντων η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις απορρίψεις είναι ανήθικο που δεν είναι λογογιάται τη βιωσιμότητα της ε, κοινή πολιτικής αλλία. Το μόνο πράγμα που δουλεύει στην πολιτική αυτή και που δουλεύει αντίστροφα από τη βάση προς το κέντρο, προς τα πάνω είναι η η η προστασία του περιβάλλοντος και η επιβολή προστήμων ε, και η έλεγχη για ό, σε όλα τα κράτη-μέλη βεβαίως υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις αλλά τα πράγματα εφαρμόζονται διαφορετικά ε, εδώ λοιπόν δουλεύει αντίστροφα το σύστημα. Αν λειτουργούσε από το κέντρο προς τη βάση, ίσως πιο ήταν, ήταν πιο ενιαία, ενιαία τα πρόστιμα ή οι, οι ποινές. Λοιπόν κύριε Μποργ προσέξτε και το θέμα αυτό αν δεν θέλετε να υπάρχει τεράστια ε, ανησυχία ή έως και αναταραχή στον τομέα. Ε, Ισλανδία τώρα και αλλιευτική συνεργασία κτλ. Ναι, ξέρω ότι συζητούμε για νέες χώρες και προ, προς χώρες και λοιπά Αλλά ε, για την Ισλανδία συγκεκριμένα σχετικά με τις συμφωνίες τι προβλέπετε Κύριε Στήλερ σα δώσω το λόγο. Αλλά επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι έχουμε πολλού προσκεκλημένου. Ότι εδώ έχουμε για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Σα παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν μπορώ να ελέγξω το, το, το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Βοηθήστε με και ελέγξτε τον χρόνο τον οποίο έχετε στη διάθεσή σα εσεί. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαστε εδώ πιο σύντομοι. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή ε, και τον Επίτροπο για το γεγονό ότι αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα προβλήματα. Μιλήσατε για την ε, ε, αποκέντρωση στην κοινή αλευτική πολιτική. Συμφωνούμε και ελπίζουμε να εξακολουθήσει αυτή η τάση. Αλλά για να δούμε. Γιατί απέτυχε η ε, υπεραλιευτική υπεραλίευση, μικρή, μικρός βαθμός συμμόρφωσης και εδώ είναι θέματα τα οποία και έχουμε και αυτή την έκθεση του συνάδελφου Ρωμέβα. Ελπίζω οι συνάδελφοι να ενδιαφερθούν για όλα αυτά τα ζητήματα. Η κυρία Ντόιλ μίλησε για ισότιμη μεταχείριση. Βεβαίω. αυτό πρέπει το δούμε και στον κανονισμό για τη συμμόρφωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι προ την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία γιατί όσο τον ε, πιο γρήγορα δράσουμε, τόσο καλύτερο. Σε σχέση με αυτά που ο κύριο ε, Στίβενσον για, το, για του καρχαρίε. Ε, ναι, καλή πρόταση επιτροπή, εδώ και καιρό τι θέλαμε. Θα, θέλω, θα ήθελα επίση να ληφθεί και κάποια δράση όσον αφορά ε, ε, ε τα, θαλασσοπούλια όπου εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά ε, και ε, εδώ πρέπει να πούμε ότι απειλούνται ιδιαίτερα ορισμένα είδη και πραγματικά αυτό είναι ένδειξη όταν πεθαίνουν τα θαλασσοπούλια καταλαβαίνετε τι γίνεται με τα αποθέματα ε, εν συντομία, μιλήσατε για τις διεθνείς υποχρεώσεις. Ο κύριος Στίβενσον επίσης ε, μίλησε ε, για, το, για, το, για, τα, για τα ψάρια και το πού τα βρίσκουμε. Κοιτάξτε, εδώ ε, ε, ακούσαμε τι γίνεται ε, όσον αφορά τους πρόσφυγες από τη Βιρμανία, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αποτελούν αντικείμενο δουλεία για να εργαστούν στους, ε, στους τόλους, να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Όλα αυτά συνδέονται και πολύ συχνά δεν δίνουμε την προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό. Εδώ μιλάμε για, εμπόριο ανθρώπων και τελικά αυτά τα ψάρια θα καταλήξουν στις δικές μας αγορές. Άρα όλα συνδέονται μεταξύ τους και όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ κύριο Γκλαβάκης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε που είστε σήμερα εδώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Από τις πολλές ερωτήσεις θα κρατήσω μόνο δύο. Ε, ε, η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω, στα πέντε χρόνια που είμαι εδώ κύριε Επίτροπε, έχω καταλάβει ένα πράγμα. Νόμους, διατάξεις, αποφάσεις έχουμε. Εκεί που υστερούμε είναι στην τήρηση των νόμων τι σκέφτεστε να κάνετε ώστε να έχουμε μια καλύτερη εφαρμογή των νόμων και των αποφάσεων. Θα αναφέρω σαν σύντομο παράδειγμα το θέμα του τόνου που δύο χρονιές υπεραλλιεύεται από κάποια κράτη, στο μέσο της χρονιάς σταματάει η αλλίευση του τόνου και αυτό επειδή δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Το ερώτημα είναι επομένως τι πρέπει να κάνετε όχι για να ψηφίσουμε καινούριους νόμους, να πάρουμε καινούριε αποφάσεις, αλλά να τηρηθούν οι υπάρχουσες που είναι αρκετές και επαρκείς το δεύτερο και τελειώνω κυρία πρόεδρε είναι το εξής λέμε ότι μειώνονται τα εχθειοποθέματα λέμε ότι τα επόμενα χρόνια ακόμη περισσότερα αλλιεύματα θα ζητιούνται από τους καταναλωτές ως μια άριστη τροφή για να την ε, καταναλώσουν. Ως εκ τούτου, εάν πρέπει να σταματήσουμε την υπεραιτέρω υπεραλίευση, πρέπει να ενισχύσουμε την, τα ηχθειοτροφία. Τι σκέφτεστε να κάνετε για περαιτέρω ενίσχυση των ιχθυοτροφίων ώστε περισσότερα ψάρια να παράγονται σε αυτά και λιγότερα να λιεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κλαβάκη. Κύριο Καπούλα, μην μου πείτε ότι θα είστε σύντομο, απλά και μου το πείτε να είστε σύντομο. Eh, κύριε... Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση του εγγράφου της Κομισιόν για το μέλλον της ΚΑΛΠ. Συμφωνώ ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά εργαλεία και αρχές, αν και πολλές φορές τα αποτελέσματα, η λειτουργία τους δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Ορισμένες από τις προτάσεις σας είναι σαφώς σωστές, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να διατηρήσουμε βιώσιμα επίπεδα ενώ ταυτόχρονα ε, ενώ ταυτόχρονα θα κρατάμε και τα επίπεδα της απασχόλησης. Και μιλάω ιδιαίτερα για τις μικρότερες και πιο απομακρυσμένες αλλιευτικές κοινότητες. η σημερινή αλληλείς είναι αυτή που θα χρειαστεί να πληρώσουν το τίμημα για τη βιώσιμη, που χρειάστηκε ήδη να πληρώσουν το τίμημα για τη βιώσιμη αλληλεία, αλλά με τι θα αποζημιωθούν και οι επόμενες γενιές θα αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό στην παρουσίασή σας αλλά και στις προτάσεις της Κομισιόν να υπάρχει μια περισσότερη εξισορρόπηση. Ευχαριστούμε κύριος Κίντερμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, εν μία ερώτηση έχω μιλήσει, μιλήσατε αν κατάλαβα καλά για ανάγκη απλούστευσης της πολιτικής τι εννοείται με τον όρο απλούστευση απλούστευση για την Κομισιόν απλούστευση για τα κράτη-μέλη ή σε τελευταία ανάλυση απλούστευση για αυτούς για τους αλλοίς και πως το φαντάζεστε εσείς θέλετε απλούστευση της νομοθεσίας ή απλούστευση της εφαρμογής των νόμων. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, θα πάρετε το λόγο να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό σιωνός για το μέλλον για τις μελλοντικέ συζητήσεις που θα κάνουμε για το μέλλον της κοινή πολιτικής αλίας. Είπα στην παρέμβασή μου, το λέμε και στην πράσινη βίβλο, αυτό που θα προτείνουμε, ότι θα κάνουμε τα πάντα, ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που δεν θα συζητήσουμε ή ενδεχομένως θα αναθεωρήσουμε άκουσα ορισμένα σχόλια για το ότι πρέπει να διατηρηθεί μια κάποια σχετική σταθερότητα. Διαφορετικά αν διαταράξουμε τα πάντα ε, δεν θα πετύχουμε τίποτε. Κοιτάξτε η θέση της Κομισιόν είναι ότι δεν θέλει να προδικάσει τίποτα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα πάντα. Ένα είναι μοναχά το θέμα το οποίο δεν μπορούμε να θίξουμε το γεγονός ότι εδώ πρόκειται για κοινή πολιτική δηλαδή για πολιτική η οποία είναι ενσωματωμένη στις συνθήκες και στην πολιτική της Λισαβόνας ε, να καταργήσουμε κοινή πολιτική ε, σημαίνει να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη άρα αυτό δεν γίνεται αλλά η μορφή που θα πρέπει να πάρει η κοινή αυτή πολιτική είναι αντικείμενο συζήτησης το κατά πώ θα διατηρήσουμε τα τάξ και τις ποσοστώσεις όσα έχουν το κατά πώ θα τα καταργήσουμε τελείως και θα την καταστήσουμε από κάτι καλύτερο το κατά πόσο θα τα συνδυάσουμε με άλλα μέτρα όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν για αυτό θα κάνουμε λοιπόν τους επόμενους μήνες. Θα ασχοληθούμε με τα πάντα και θα συζητήσουμε όλα τα πιθανά σενάρια. Και θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω μερικές τουλάχιστον από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Πρώτον, πρώτη ερώτηση, ε, πόσο χρόνο θα διαρκέσουν οι διαφουλεύσεις μετά την ε, δημοσίευση πράσινης βίβλου. Κοιτάξτε, ελπίζουμε ότι μια πρώτη άτυπη συζήτηση στο Συμβούλιο θα γίνει τέλος Απριλίου ή Μάιο στο Συμβούλιο και μετά έχουμε κατά νου γύρω στους έξι μήνες διάρκεια μέχρι το τέλος χρονιάς δηλαδή ο, για τη δημόσια διαβούλευση με όλες τις κατηγορίες ενδιαφερομένων όχι απλώς τις συνήθεις κατηγορίες αλλά όλους, όλο το κοινό όλη την κοινή γνώμη χρειαζόμαστε όλους τους ε, τομείς πρέπει να τους εμπλέξουμε στις συζητήσεις που θα γίνουν ελπίζω μετά από αυτές τις ευρύτατες συζητήσεις να καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα στη διάρκεια του 2010 ούτως ώστε να φτιάξουμε υποβάλουμε και μια νέα και μια, την... μια πρόταση για τη νέα πολιτική αλίας ε, η οποία θα έρθει σε εσά και στο, θα πάει στο Συμβούλιο και ελπίζουμε η νέα αυτή πολιτική να εγκριθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης αν τα πράγματα ε, πάνε καλά με τις ενδείκτες της Λαβώνας μέχρι το τέλος του 2012. Υπάρχει χρόνος με άλλα λόγια. Γι' αυτό ξεκινούμε τις συζητήσεις αρκετά νωρίς για να έχουμε ε, συζητήσεις ως το δυνατόν πιο ευρείες και ανοιχτές. Τώρα για την κυρία Φράγκα και τις ερωτήσεις της για τα τάξη και τις που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι βεβαίως θα πρέπει να καθίσουμε να δούμε αν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Θα θέλαμε να γίνει συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση της αλληλευτικής προσπάθειας. Ε, θα πρέπει να δούμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις θα πιστεύουμε ότι ο κλάδος πρέπει να συμμετέχει πιο πολύ και να αναλάβει περισσότερες ευθύνες η μικροδιαχείριση να γίνεται από τον ίδιο τον κλάδο να μην χρειάζεται να πάμε κάθε φορά στο Συμβουλίο για να πάρθουν αποφάσεις για την καθημερινότητα για τις καθημερινές ενέργειες στον τομέα της αλίας αλλά οι βασικές πολιτικές ε, κατευθύνσεις θα πρέπει να αποφασίζονται σε ψηλότερο επίπεδο και θα μπορούσαν κάλλιστα να αποφασίζονται και σε εθνικό επίπεδο. Τώρα για την εξωτερική πολιτική που ανέφερε η κυρία Φράγκα για τις διμερείς συμφωνίες και αυτά θα καλυφθούν στην πράσινη βίβλο αλλά αναμένουμε οι συζητήσεις να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο το ώστε να δούμε κατά πόσον υπάρχει μέλλον για τις συμφωνίες αυτές κατά πόσον πρέπει να αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους ή κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως κατεύθυνση. Αυτά είναι βασικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε προβλήματα όπως ξέρετε με το ο, με τις συμφωνίες αυτές ε, με τις τρίτες χώρες για τις εταιρικές σχέσεις ε, θα πρέπει να βρούμε μια καλή λύση αν θέλουμε να συνεχιστούν οι συμφωνίες αυτές στο μέλλον και αν θέλουμε να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο ούτω ώστε οι τρίτες χώρες, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους στο θέμα της Ελίας. As well. Um, we ε, ε, για το άρθρο 47 για την εραστιχνική αλληλεία πράγματι θα ελπίζουμε να αναθεωρήσουμε τις διατάξεις του άρθρου αυτού και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση εμείς και εσείς ως Επιτροπή για να μπορέσουμε τελικά να έχουμε μια νομοθετική διάταξη εκεί ε, η οποία να αναφέρεται μοναχά στην εραστεχνική αλληλεία η οποία δημιουργεί πιέσεις για τους ελευτικούς πόρους αντίστοιχου μεγέθους όπως οι πιέσεις των επαγγελματιών αλλιέων. Όπως είπα και πριν Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι πόροι τους οποίους προσπαθούμε να ξανααναπτύξουμε και μιλάμε για την αλληλεία από σκάφη. Προσπαθούμε να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή η οποία να μας προ... να... Ναι, επι ανάλογα με το στόχο που επιδιώκουμε η οποία να ε, χωρίζει την εραστεχνική αλία που δεν ενοχλεί από αυτήν η οποία είναι έως και επικίνδυνη. Τώρα, <clears throat> είναι γεγονός ότι ο οριζόντιος κανονισμός τους τελευταίους τις τελευταίες εβδομάδες περνώντας από το, στη συζήτησή του για, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ε, απέκτησε μια κάποια ορμή και γι' αυτό και εμείς ε, ασχοληθήκαμε την οριζόντια οδηγία γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά θα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί για τις οικολογικές ετικέτες αυτές πιστεύουμε ότι το σύστημα αυτό ε, θα ήταν καλύτερο αν είχαμε μία ε, ετικέτα, ο καθένας είχε το δικό του σύστημα. Τέλος πάντων ξέρουμε ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα και υπάρχουν ιδιαιτερότητες ελπίζουμε να μπορούμε να κάνουμε να διαχωρίσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες στην, στις οριζόντιες νομοθετικές πράξεις ίσως μέσω, ή, ίσως μέσω ενός παραρτήματος με, ή με κάποιο άλλο τρόπο και θα κάνουμε την ε, συζήτηση και τη μελέτη αυτή και αν τελικά αποφασιστεί ε, η πρότασή μας δεν γίνει αποδεκτή ε, για την αλία μες στο γενικό πλαίσιο θα συνεχίσουμε με ειδικό eco-labeling για την αλία όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση τώρα αυτό που είπε ο κύριος Κασάκα για τις περιφερειακές περιοχές τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Βεβαίως θα ληφθούν αυτές υπόψη στο, στην, ε, στο διαχωρισμό σε περιφέρειες των υδάτων και όπως είπα και πριν θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε την μικροδιαχείριση, την εφαρμογή των κανόνων σε κάποιες στις συγκεκριμένες περιφέρειες εφόσον αυτές βέβαια συνάδουν με το γενικό πλαίσιο στην ίδια την περιφέρεια. αυτού του είδους στην αποκέντρωση θέλουμε να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Νομίζω ότι τελικά άμεσα ή έμεσα έχω απαντήσει σε πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Χάτστον για την κοινή πολιτική αλίας τώρα για την ίση πρόσβαση στα ύδατα και στους πόρους όντως η αρχή αυτή ισχύει αλλά σήμερα όλα εξαρτώνται από το θέμα της σχετικής σταθερότητας αν από Μακριθούμε λοιπόν από την αρχή της σχετικής σταθερότητας τότε θα πρέπει να βρούμε ένα εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης δίκαιο κατά την εφαρμογή του. Πριν πάρουμε λοιπόν οποιασδήποτε αποφάσεις αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τώρα για τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια πιστεύουμε ότι τα συμβούλια αυτά πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες κατά πόσον είναι ο τέλειος ή ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε τα συμβούλια αυτά δεν το ξέρω θα πρέπει να το δούμε και αυτό σίγουρα όμως πιστεύουμε ότι ο, η ρόλος και συμβουλευτικός ρόλος των συμβουλίων αυτών είναι πολύ σημαντικός και πιστεύουμε και ότι και άλλες ε, άλλοι φορείς όπως παραδείγματος χάρη είναι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να αναλάβουν παραπάνω ευθύνε, γιατί αυτοί είναι οι αλληλείς οι οποίοι δουλεύουν στον τομέα και οι οποίοι πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους και να σεβαστούν κάποιες ευθύνες. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα ε, μας οδηγήσουν σε καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση. Για αυτά που είπε ο κ. Στίβενσον για την αποτυχία, το είπε και ο κ. Σάλιστερ αυτό, για την αποτυχία της κοινή πολιτικής. Αλλά συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θα ήμουν τόσο αρνητικός, γιατί, διότι εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην επιτύχαμε τους στόχους που επιδιώκαμε. Γιατί ακριβώς προχώρησε τόσο πολύ η αλληλεία αυτή καθεαυτή οι τεχνολογικές πρόοδοι παραδείγματος χάρη που ξεπέρασαν αυτού τους στόχους οι παλιοί κανόνες δεν μπορούσαν να προβλέψουν τη μεγάλη πρόοδο που θα γινόταν στον κλάδο και όπως είπαν και κάποιοι ομιλητές το τότε παλιά όταν φτιάχναμε την κοινή πολιτική αλληλεία το πρόβλημα ήταν ο έλεγχος και σωστή εφαρμογή. Μπορεί κανείς να φτιάξει μια κοινή πολιτική αλληλεία τέλεια ή όχι τόσο τέλεια άμα όμως δεν υπάρχουν σωστοί έλεγχοι και εφαρμογή τότε δεν δουλεύει τίποτα. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολιτική αλληλείας πολύ λιγότερο μικρότερης εμβέλειας από αυτή που έχουμε. Αν είχαμε λοιπόν λιγότερο φιλόδοξους στόχους θα τους είχαμε επιτύχει. Όμως ε, εμείς ε, πήγαμε πιο πέρα ε, είχαμε μακρόπνους και φιλόδοξους στόχους ε, οι, βεβαίως οι έλεγχοι δεν δουλεύουν σωστά ε, και πρέπει να αναθεωρηθούν Κα, καταλαβαίνω ε, από την άλλη μεριά ότι ό,τι και να κάνουμε αν οι έλεγχοι δεν πάνε καλά δεν γίνουν αποδεκτό, αν δεν γίνει αποδεκτό το σύστημα των ελέγχων τότε κάποιος πάντα θα υπάρχει που θα γκρινιάζει. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και τη συζήτηση για το σύστημα των ελέγχων. Μόνο αν έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτά και άλλα πράγματα στην κοινή πολιτική αλίας. Τώρα, Τώρα για την ηχθειοκαλλιέργεια. Έχουμε και γι' αυτό προβλέψει μια πράσινη βίβλο που θα βγει στις αρχές Απριλίου και τη βλέπουμε παραλίλω με την συζητήση της μεταρρύθμισης της ΚΑΛΠ. Θα μπορούσαν και να συγχωνευτούν αλλά έχει νόημα και να παραμείνουν χωριστές για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το μέλλον της ηχθειοκαλλιέργειας χωριστά. Δεν είναι θέμα κοινή πολιτικής και άρα η, το, η δικαιοδοσία μας είναι πολύ μικρότερη. Παρ' αυτά ελπίζουμε να μπορέσουμε να ε, εκλογικεύσουμε τον αριθμό των ε, κανονισμών που ισχύουν και που προκαλούν σύγχυση. Μερικές, ε, μερικοί από αυτούς τους κανονισμούς αφορούν την υγεία, όχι άμεσα την ηχθειοκαλλιέργεια, αλλά απλώ αναφέρεται. Ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να γίνει και μια συζήτηση για την ηχθειοκαλλιέργεια, ίσως και ακρόαση, στο Συμβούλιο. Και επίσης στο Συμβούλιο που να εγκρίνει τα σχετικά συμπεράσματα πριν τα τέλη του χρόνου. Τώρα για τις απορρίψεις, ναι βεβαίως δεν βασιζόμαστε συγκεκριμένα στις απορρίψεις στη συζήτηση αυτή της πρασίνης βίβλου, αλλά οι απορρίψεις κατ' εμάς πρέπει να είναι, η κατάργηση των απορρίψεων, ε, από τους τελικούς μας στόχους αλλά όχι με μορφή απαγόρευσης αλλά ένας από τους τελικούς στόχους οποιασδήποτε μεταρρύθμισης της ΚΑΛΠ. Αυτό είναι σαφές. Δεν αναφέρουμε συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχουμε αυτό γιατί αυτό εξαρτάται και από τη γενική μορφή που θα πάρει η μεταρρύθμιση αλλά σίγουρα είναι ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να, να έχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο είχε αποφασίσει την απαγόρευση του high grading που είναι ένα είδος απόρριψης που κάνουν οι αλληλείς όπως είπε και η κυρία Ντόιλ είναι υποχρεωμένοι να απορρίπτουν ορισμένα είδη ψαριών για να μην κατηγορηθούν ως παραβάτες του νόμου. Ορισμένοι τα απορρίπτουν ψόφια στη θάλασσα απλώς και μόνο γιατί χρειάζονται περισσότερο χώρο για να αποθηκεύσουν εκεί καλύτερης ποιότητας ψάρια. Αυτό είναι το upgrading. Και υπάρχουν επίσης συμβαίνουν και άλλα με τις απορρίψεις όπου ορισμένοι αλληλείς απορρίπτουν ψάρια απλώς γιατί τους βολεύει περισσότερο χωρίς να ξέρουμε ακριβώς γιατί. Αυτά που είπε ο κύριος Ρωμέβα για την μείωση του αριθμού των αλλιευτικών πηλιαρίων. Έχουμε προτείνει μία δέσμη μέτρων για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στους αλείς ή στις χώρες μέλη για να κάνουν μία αναδιάρθρωση των στόλων τους όποτε θεωρούν ότι υπάρχει υπάρχουν υπερβολικά πολλά αλληλευτικά πλοιάρια. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι μερικά τμήματα του αλληλευτικού μας στόχου είναι άχρηστα. Όχι όλος ο στόλος βέβαια, αλλά σε πολλά σημεία υπάρχει υπερβολικός αριθμός και θέλουμε να δούμε ποια είναι τα καλύτερα κίνητρα όπως μεγαλύτερες δυνατότητες για το αλλιευτικό, για καλύτερη χρησιμοποίηση του αλλιευτικού ταμείου αλλά δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα όλα αυτά όπως τουλάχιστον περιμέναμε και ελπίζουμε να καταλάβουν οι χώρες μέλη και οι αλληλείς οι ίδιοι περισσότερο ότι κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα σύντομα και ως προς αυτόν τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό πλειάριων Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο τότε θα συνεχίσει ο πειρασμός όλο και περισσότερων αλλιεύσεων και αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα όταν θέλουμε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Είναι λοιπόν ζωτικό να το αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα έχει γίνει κάποια πρόοδος αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, πολύ περισσότερα πράγματα. Και είναι και αυτό ένα από τα τμήματα της αερομεταρρύθμισης της ΚΑΛΠ. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Α, μιλήσατε και για το σχέδιο δράσης των καρχαριών και άλλοι για τα θαλασσοπούλια αρχίζουμε να το εξετάζουμε, ακόμη αρχίζουμε και όταν έχουμε κάτι να σας πούμε θα σας το υποβάλουμε δεόντως και είναι ευθέτω χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε τώρα γιατί ακόμη δεν, έχουμε καταλήξει. Θέλουμε πρώτα να δούμε πώς είναι η κατάσταση και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Για τους πρόσφυγες από τη Βυρμανία θα το εξετάσουμε να δούμε αν όντως υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και τότε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τη μεριά μας. Βέβαια δεν είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι. Εγώ είμαι αρμόδιος μόνο για την αλληλεία, αλλά θα το δούμε. Ο κύριος Γκλαβάκης μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει πιο, αυστηρή, πιο αυστηρός των κανόνων. Αυτό το αρχίσαμε ήδη να το συζητάμε για το νέο κανονισμό εφαρμογή των ελέγχων που ελπίζουμε να εγκριθεί πριν λήξει το έτος αλλά ελπίζουμε επίσης να μην καταλήξουμε τελικά σε αποδυνάμωση των ισχυών των κανόνων από λόγω πιέσεων που θα ασκηθούν από διάφορους από διάφορες πλευρές γιατί τότε θα καταλήξουμε σε μια καλή μεν ίσως μεταρρύθμιση αλλά που δεν θα εφαρμόζεται. Αυτό δεν θέλουμε να γίνει και γι' αυτό είχα μιλήσει και για την ερασιτεχνική αλληλεία. Ήταν τμήμα των προτάσεων για τον έλεγχο, αλλά φυσικά, φυσικά δεν, θα, δεν έχουμε στόχο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύουν οι πραγματικοί ερασιτέχνες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για πραγματικά ερασιτέχνες αλλά για και καλυμμένη εμπορική δραστηριότητα και άσκηση πιέσεων ε, που καταλήγουν σε μείωση των αποθεμάτων και τελικά θα βλαφτούν περισσότερο από τους άλλους και, και οι ερασιτέχνες ψαράδες. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και να βρούμε λύσεις εξισορροπημένες και λογικές. Για τις μικρές αλλιευτικές κοινότητες τώρα, ναι πράγματι, το είπε ο κύριος Καπούλας, φυσικά πρέπει να το δούμε και αυτό προσεκτικά, αλλά και αυτό εξαρτάται από το είδος διαχείρισης που θα εφαρμοστεί αν ας πούμε όπως είπε η κυρία Φράγα μιλήσουμε για τις μεταφορές ή τις πωλήσει ποσοστώσεων αν υπάρξει ένα σύστημα που να συμπεριλαμβάνει και αυτό το ITQ, δηλαδή τις μεταφερόμενες ποσοστώσεις, τότε θα πρέπει ιδιαίτερη μέρη να δοθεί για τις μικρές αλληλευτικές κοινότητες στις μικρές ελευθερικές κοινότητες που μπορεί να υποφέρουν από την εφαρμογή του συστήματος. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι είναι το καλύτερο. Τέλος, αυτά που είπε ο κύριος Κίντερμαν για την απλοποίηση. Ελπίζω η απλοποίηση να τονίσει, να βασιστεί στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Να φύγουμε δηλαδή από τη μικροδιαχείριση και να πάμε σε πολύ ευρύτερο επίπεδο διαχείρισης αφήνοντας την πρώτη, τη μικροδιαχείριση δηλαδή, στους ε, άμεσα ενδιαφερόμενους. Αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει μεγαλύτερη απλοποίηση. Τελικά όμως η ουσία είναι το σύστημα που θα εφαρμοστεί να είναι κατανοητό ακριβώς από τους ενδιαφερόμενους που θα χρειαστεί να το λειτουργήσουν που είναι, ελπίζουμε να είναι, και αυτή αναπόσπαστο τμήμα στην ίδια τη διαδικασία της διατύπωσης των κανόνων που θα χρειαστεί να εφαρμόσουν. Ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Βέβαια και αύριο ξέρω ότι θα συζητήσετε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Α, α την Ισλανδία, την Ισλανδία, ναι. Την Ισλανδία, πού την έχω την Ισλανδία. Α, ναι, εδώ, λοιπόν. Ναι, αυτά που είπε η κυρία Ντόιλ για την Ισλανδία. Ναι, ναι, ναι, τα έχω εδώ. Λοιπόν, εδώ. Αν η Ισλανδία αποφασίσει να ζητήσει ένταξή της στην Ένωση, που είναι κάτι που έχει δικαίωμα να το κάνει και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, εκείνη μόνη της θα δει αν θέλει να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Αλλά αν αποφασίσει να υποβάλει αίτηση, εμείς θα πρέπει να συζητήσουμε με τις αρχές της Ισλανδίας ποιο σύστημα διαχείρισης της αλίας εφαρμόζουν, της αλίας τους, έτσι ώστε η κάλπ να εφαρμόζεται με τρόπο που να μην δημιουργεί, να μην ζημιώνει και τους Ισλανδούς αλληλείς. Αυτό βέβαια θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις, στις συνταξιακές διαπραγματεύσεις όπου πάντοτε για όλες τις χώρες λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Το κάναμε για όλες τις χώρες. Όταν καθορίσαμε ας πούμε την ζώνη των 25 μιλίων υπάρχουν τρόποι που μπορούμε μέσα με τους κανόνες της ΚΑΛΠ να λάβουμε υπόψη μας και τις ιδιαιτερότητες ορισμένων χωρών αλλά όχι opt-out από την πολιτική αυτή γενικότερα. Είναι τμήμα του κεκτημένου και καμία χώρα μέλος ή υποψήφια χώρα μέλος δεν μπορεί να ζητήσει γενική εξαίρεση από την πολιτική αυτή. Από καμία κοινή πολιτική. Αυτό αποκλείεται. Εάν όμως οι αρχές της Ισλανδίας είναι διατεθειμένες να συζητήσουν με ποιον τρόπο η ΚΑΛΠ θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις πραγματικότητες της Ισλανδίας, τότε φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Κάτι άλλο. Η ίδια η μεταρρύθμιση της που θα μπορούσε να κινηθεί προς την κατεύθυνση να εμπνευστεί από τη διαχείριση που εφαρμόζουν ορισμένες βόρειες χώρες όπως η Νορβηγία και η Ισλανδία. Μπορεί η ΚΑΛΠ να καταλήξει τελικά να εφαρμόσει ένα σύστημα που να είναι πιο κοντά σε αυτό που εφαρμόζουν ορισμένες τέτοιες χώρες. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουμε και να το εξετάσουμε. Τέλος, επειδή η Ισλανδία είναι εταίρος μας στην Αλία όπως και η Νορβηγία, την καλέσαμε, τη ζητήσαμε να ορίσει έναν εκπρόσωπο ανεξαρτήτως από το αν θα υποβάλει αίτηση ή όχι, να ορίσει εκπρόσωπο στις συζητήσεις για την μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ ώστε και μόνοι τους να μπορέσουν να δουν να αποτελέσουν τμήμα της ομάδας που τελικά θα διαμορφώσει μία ριζική ελπίζω μεταρρύθμιση μίας βασικής κοινής πολιτικής μας. Τελεία. Σας ευχαριστώ. Νομίζω Νομίζω ότι η παρέμβαση αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Ε, συναρπαστική συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το έργο μας. Κοιτάξτε, πραγματικά όσον αφορά το χρόνο μας πιέζει ιδιαίτερα, δεν σας το κρύβω. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε τρεις ενότητες με τρεις ε, ομιλητές κάθε μία. Ξεκινώ λοιπόν με, με την πρώτη ενότητα εμπειρογνωμόνων. Οι τρεις πρώτοι εμπειρογνώμονες είναι ο κύριος Άντερσον, που προέρχεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βόρειας Θάλασσας, ο πρόεδρος, ο κύριος Σου, ε, που είναι ε, σύμβουλος του Υπουργού Τροφίμων Γεωργίας και Ελίας της Δανίας και τον κύριο Πούλεν που ε, είναι διευθυντής ε, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Τροφίμων και Υπέθρου του Ηνωμένου Βασιλείου. Κοιτάξτε, στον καθένα σας θα δώσω 10 λεπτά. Ε, κοιτάξτε, στη συνέχεια θα είμαι αναγκασμένη να σας διακόψω, γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να τελειώσουμε σε 6.30. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περισσότερο. Θα έχουμε λοιπόν μετά από κάθε ενότητα 10 λεπτά όπου θα μπορούν να θέσουν ερωτήσεις και να δεχθούν απαντήσεις από εσά τα μέλη της Επιτροπής. Να δώσουμε πρώτο λόγο στον κύριο Άντερσον. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω κάθε προσπάθεια να μιλήσω λιγότερο από 10 λεπτά, γιατί πολλά από τα οποία, ε, τα οποία ήθελα να θίξω αναφέρθηκαν στην προηγούμενη συζήτηση. Λοιπόν, Αρχίζω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που με κάλεσε εδώ και μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Βρισκόμαστε βεβαίως σε ένα πρώιμο στάδιο όσον αφορά αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης ε, της ε, κοινή ε, πολιτικής αλίας και λόγω του γεγονότος αυτού το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στο οποίο είμαι πρόεδρος, δεν έχει ακόμα υποβάλει επίσημα την γνωμοδότησή του για το θέμα αυτό. Πάντως θα το πράξουμε στη συνέχεια, μέσα στο χρόνο. Αυτά τα θα σας πω λοιπόν σήμερα αφορούν τη δική μου ερμηνεία όπως, όπως βλέπω εγώ δηλαδή την άποψη του Συμβουλίου μου, αλλά θα σας μεταφέρω και τη δική μου άποψη. Για να δούμε τα αποτελέσματα ε, της ε, προηγούμενης αναθεώρησης. Όσον αφορά την καλή διακυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Την καλή διακυβέρνηση ε, η οποία κατέληξε ε, ακριβώς στη δημιουργία αυτών των περιφερειακών γραμματικών συμβουλίων. Κατά τη διάρκεια του προβληματισμού ακούστηκαν απόψει για το ότι δεν θα πρέπει μόνο να είναι γνωμοδοτικά, αλλά να είναι και διαχειριστικά τα συμβούλια αυτά. Στη δική μου περίπτωση, πάνω από τέσσερα χρόνια ε, έχουμε την εμπειρία του γνωμοδοτικού συμβουλίου και πιστεύω ότι ήταν το σωστό βήμα αυτό που, ε, που ελήφθη τότε. Και πραγματικά ελπίζω να βοηθήσαμε και να συμβάλαμε για στην βελτίωση της κοινή πολιτικής αλίας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε τα... Να πούμε κάτι το οποίο ε, είναι, είναι στοιχειώδες. Δηλαδή, οι αποφάσεις πρέπει στο σωστό επίπεδο. Αυτό το είπε και ο Επίτροπος Μπόρκ στην ε, προηγούμενη του παρέμβαση σήμερα. Δεν είναι δυνατόν σε επίπεδο υπουργών να γίνονται όλε αυτέ οι λεπτομερεί συζητήσει. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα σύστημα όπου οι αποφάσει λαμβάνονται στο σωστό επίπεδο και βεβαίω το ένα επίπεδο είναι το περιφερειακό επίπεδο, άλλο το εθνικό, αλλά και το τοπικό. Πώ θα τα οργανώσουμε όλα αυτά. Αυτό το, αφήνω το ερώτημα αυτό να απαντηθεί από άλλους ομιλητές. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ε, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια με την εφιστάμενη τους δομή δεν μπορούν να γίνουν διαχειριστικοί φορείς. Η οργάνωσή μας στηρίζεται το γεγονό ότι είμαστε γνωμοδοτικά συμβούλια, όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε εθελοντική Βάση. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε μια άλλη δομή σε περιφερειακό επίπεδο που να ε, επιτρέπει τη μετατροπή των συμβουλίων αυτών και σε διαχειριστικά. Αυτό όμως, όπως σας είπα, θα το αφήσω στην άκρη. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν λύσεις που θα προταθούν. Αρκεί να κοιτάξουμε πέραν του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε. Όπου υπάρχει ένα είδος κοινή ε, πολιτικής αλίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο, και στη συνέχεια υπάρχουν οι περιφερειακές μονάδες διαχείρισης. Άρα λοιπόν έχουμε παραδείγματα καλής πρακτικής από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Όσον αφορά το θέμα του ελέγχου, θέμα το οποίο προκύπτει να συζητάμε την κοινή πολιτική ελίας. Εδώ βεβαίω συζητάμε το θέμα των πόρων ε, κτλ. Το θέμα του ελέγχου όμω αποτελεί σημαντικό τμήμα τη κοινή πολιτική αλεία. Και στο δικό μου γνωμοτικό συμβούλιο, με τις, ε, τον κοινοτικό φορέα ελέγχου της Αλίας διοργανώνουμε ε, διασκέψεις για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και, συζη... και ανταλλάσσουν απόψη το θέμα του ελέγχου και τη συμμόρφωση. Αυτή η διάσκεψη που έγινε πριν από ένα χρόνο σε εμά ήταν πάρα πολύ σημαντική ε, και μα βοήθησε να έχουμε πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων. Ε, ε, έχουμε κάνει τα σωστά βήματα προ σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα. Και άλλα, και άλλα. Για να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και να συμμορφωνόμαστε με τι υποχρεώσει. Διότι εάν οι εμπλεκόμενοι, οι αλλοί σε αυτή την περίπτωση δεν κατανοούν τους κανόνες ή δεν δέχονται τους κανόνες αυτούς ή δεν μπορούν να, τους, ε, ε, να συμμορφωθούν τους κανόνες αυτούς για πρακτικούς λόγους, ε, τότε θα έχουμε παραβάσεις. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων ξεκινά με το διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό με τσολίζει βασικά. Αυτό τη στιγμή θέσπιση των κανόνων. Πρέπει ευθύ εξ αρχή να συμμετέχουν οι αλληλεί, έτσι ώστε να, να καταλάβουν πλήρω το τι γίνεται, του λόγου του οποίου γίνεται και να συμβάλλουν και εκείνοι με τι δικέ του ιδέε. Από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Με τη συμμετοχή όλων. Εάν δεν το πράξουμε, τότε δεν έχει νόημα να έχουμε περισσότερους επιθεωρητές και περισσότερους ελέγχους. Αυτό που απαιτείται είναι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τώρα, να κάνω ορισμένα σχόλια για τους πόρους. Και κάτι το οποίο αναφέρθηκε και νωρίτερα. Το θέμα των απορρίψεων. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαράδεκτο. Από κάθε άποψη. Από όλους. Να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα διαχείρισης που δημιουργεί απορρίψει. Αυτό βεβαίως είναι απαράδεκτο και πάψη πόρων. Ανεξάρτητα με το αν το ονομάζουμε αναβάθμιση ή έλλειψη επιλεκτικότητας ε, ε, ε στους, ε, στα, στα δίχτυα κτλ. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τις απορρίψεις. Εμείς ως πολιτικοί δεν πρέπει να έχουμε ένα, δεν πρέπει να, δημιουργούμε, να έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης που οδηγεί στη δημιουργία απορρίψεων. Αυτό πρέπει να το δούμε σήμερα. Και το μεγαλύτερο μέρος των απορρίψεων δημιουργείται από το ίδιο το σύστημα διαχείρισης. Και αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε. Mm. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω εδώ. Ε, ελπίζω να εξοικονόμησα ορισμένα λεπτά, λεπτά. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο το δώρο σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Σου. Σου. Χωρίς μικρόφωνο. I participated in the... Είχα πάει, είχα συμμετάσχει στην μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ το 1992 και το 2002 καθώς και στην εφαρμογή της το 1993. Αυτό δεν το λέω για να πενευτώ αλλά για να το γνωρίζετε. Παρακαλώ λοιπόν να μου επιτρέψετε να είμαι πολύ ομόσο στην προσέγγιση μου. Η ΚΑΛΠ έχει ως στόχο την βιωσιμότητα και την οικονομική ευμάρεια. Αλλά δεν έχει πετύχει το στόχο αυτό καθόλου. Η Δανέζικη κυβέρνηση προτείνει, και αυτό συμφωνεί απόλυτα με τη γενική και η ανάλυση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής επαναπροτείνει μάλλον μία αλλαγή στάσης και νοοτροπίας ώστε οι διακανονισμοί, οι λεπτομερείς διακανονισμοί να αντικατασταθούν από την ευθύνη του κάθε αλλιέως. Με τη χρησιμοποίηση των ιδίων πόρων βέβαια και με απλούς κανόνες, διότι στο κάτω-κάτω το κύριο θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι η αλίευση δεν θα ξεπερνάει κάποιο όγκο. Η ΚΑΛΠ διασφαλίζει το στόχο αυτό μέσω περίπου χίλιων κανόνων, των οποίων η πολυπλοκότητα είναι κατανοητή από όλους, αν και οι ίδιοι κανόνες είναι ακατανόητοι. Εμείς θέλουμε να είναι υπεύθυνος ο κάθε αλιεύς και να υποβάλει ο ίδιος τα στοιχεία για τα αλλιεύματά του. Αυτό νομίζω ότι είναι καθολικό, δίκαιο και κατανοητό. Έτοιμα για τον χρήστη των πόρων μας. Δεν θα αναφέρω πολλές λεπτομέρειες, αλλά γενικά βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι ότι η εθνική διαχείριση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του υπερβολικού όγκου των αλλιευτικών πλοιαρίων και δεύτερον αν μετρώνται τα ψάρια που φτάνουν στην ε, ακροθαλασσιά δεν μετριέται τι έχει αλλιευτεί μέσα στη θάλασσα το πρόβλημα είναι καταρχάς εθνικό και εθνική δικαιοδοσία και εθνικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουν τα κράτη. Δεύτερο πρόβλημα η ΚΑΛΠ από το 2002 και μετά ρητά ορίζει ότι το αλίευμα είναι αυτό που φτάνει στην ακροθαλασσιά. Αυτά τα ψάρια καταγράφονται και υπολογίζεται κατά πόσον συμφωνούν με την ποσόστοση και επιβάλλονται περιορισμοί και εφαρμόζονται καμιά χιλιαριά κανόνες. Η ίδια η φιλοσοφία της ΚΑΛΠ λοιπόν είναι ότι αν περιοριστεί η αλίευση για 15 μέρες, παρατηρείται μία μείωση αλλιευμάτων κατά 50%. Αυτό δεν έχει λυθεί, πώς εξηγείται, και οι αλληλείς δεν το δέχονται. Γιατί τους επιβάλλονται πρόστιμα υπερβολικά και για υπερβολικά μεγάλες περιόδους. 13 μέρες το μήνα περίπου. Είπα ότι είναι πολλά τα πλοιάρια, αλλά αυτό δεν είναι το κύριο θέμα που εξετάζω σήμερα, γιατί είναι εθνικό. Θα ήθελα μόνο να το εξηγήσω την δανέζικη εμπειρία. Οι μεταφερόμενες ποσοστώσεις δεν οδηγούν απαραίτητα σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίων ή άλλων πόρων. Από τότε που εισήχθησαν οι μεταφερόμενες ποσοστό στη Δανία έγινε, παρατηρήθηκε μια συγκέντρωση στην αλία αφρο, αφροψάρων αλλά από την άλλη μεριά μεταφέρθηκαν τα ψάρια αυξήθηκε η παράκτια αλία και όχι η αλία της ανοιχτής θαλάσσης παραπέρα βλέπετε στην προσθήκη που έχω να δώσω στη γραμματεία άμα θέλετε. Μέσω της γραμματείας μπορείτε να την πάρετε. Τώρα, εμείς θεωρούμε ότι τα μεταφερόμενα δικαιώματα σε αυτό το σύστημα ITQ θα διασφάλιζε μία προσαρμογή των μέτρων στην πραγματικότητα των αλλιέων. Δεν είναι όμως και καμία πανάκια για την καταπολέμηση του upgrading. Οι μεταφερόμενες ποσοστώσεις τελικά ελαχιστοποιούν το κεφάλαιο που χρειάζεται να κινητοποιήσει ο αλλιεύς για να κάνει τη δουλειά του. Δεν διασφαλίζει όμως την καταλληλότερη δυνατή χρήση των πόρων. Τώρα πώς θα μπορούσαν ε, να υπάρξει καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Μπορεί να υπάρξει και με βιώσιμη αλληλεία αλλά και με μεγιστοποίηση της του βιολογικού ωφέλους που μπορούμε να έχουμε από τις αλλιεύσεις. Πολύ απλοί κανόνες με τη χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν και σε άλλους τομείς. Εμείς θεωρούμε ότι οι αλληλείς πρέπει να έχουν ποσοστώσεις αλίευσης και όχι αποφόρτωσης και να παίρνουν πριμ αν δείχνουν υπευθυνότητα για τον υπολογισμό όλων τους των αλλιευμάτων. Αν γίνει αυτό τότε θα είναι πιο σωστά τα στοιχεία μας, θα έχουν βιολογικά ιδίως για τη διαχείριση των αποθεμάτων και θα γίνει επιλεκτικά η αλληλεία με βάση τα συμφέροντα των χρηστών οι οποίοι θα έχουν και καλύτερη πρόσβαση σε αγορές. Γιατί θα υπάρχει απολογισμός για όλα τα αλλιευόμενα ψάρια και ηχθείες. Πώς μπορούμε όμως να το πετύχουμε αυτό. Εμείς προτείνουμε μέσα στα πλαίσια της ΚΑΛΠ να δημιουργηθεί ένα εθελοντικό δεύτερο γενές σύστημα διαχείρισης όπου μόνοι τους οι ψαράδες να εφαρμόζουν τους ελέγχους με τον όρο να υποβάλουν σωστά στοιχεία για τις αλλιεύσεις. Μπορεί να υπάρχει και κάμερα που να τα καταγράφει τα αλλιεύματα. Αν μπορέσει να επιτευχθεί αυτό τότε θα υπάρχει δυνατότητα ενός δευτερογενούς συστήματος διαχείρισης όπου δεν αλλάζουν χέρια τα ψάρια αλλά πηγαίνουν από τον κάλαθο των αχρήστων στους ίδιους τους ψαράδες που θα μετρούν όλα τα ψάρια θα έχουμε πολύ ακριβή στοιχεία και για τα βιολογικά δεδομένα που αφορούν τα ψάρια και θα επανέλθουν τα αποθέματα. Όλοι γνωρίζουμε νομίζω ότι υπάρχει σπατάλη των αλλιευμάτων στα ενωσιακά ύδατα. Ένα εκατομμύριο τόνους το χρόνο λένε ότι απορρίπτουν. Και γενικά προβλέπεται από την ΦΑΟ και την Παγκόσμια Τράπεζα 50 εκατομμύρια να απορρίπτονται το χρόνο. Αν βρούμε μια λύση μέσα στην Ένωση για αυτό το πρόβλημα, τότε μπορεί και η Ένωση να παίξει σημαντικότερο διεθνή ρόλο στα αλλιευτικά. Την πρόταση αυτή στη Δανία έχει χρόνια που τη συζητάμε και αρχίσαμε πέρυσι ένα πρόγραμμα με το οποίο γίνεται η αλληλεία με κάμερες πάνω σε έξι πλοιάρια από το Δεκέμβριο του 2008. Έχει ήδη, δηλαδή ήδη 1,5 ολόκληρο μήνα. Αλλά μπορώ ήδη να σας πω ότι από τα πρώτα ευρήματα φαίνεται ότι τεχνικά δουλεύει το σύστημα και ότι οι αλληλείς το δέχονται ευχαρίστως. Και φαίνεται επίσης ότι τα στοιχεία από τις κάμερες είναι πολύ αξιόπιστα. Θα δούμε βέβαια πώς θα τελειώσει το πείραμα. Και τώρα θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι στην ιστοσελίδα μας που θα την δώσω στην γραμματεία προσπαθούμε να διατυπώσουμε μερικές από αυτές τις ιδέες με νομοθετικό τρόπο και ύφος καθώς και ορισμένες σκέψεις για τη διαχείριση των μεταφερομένων προσωστώσεων. Και με αυτά κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Σας κατευχαριστούμε, ήσασταν τέλειος. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πλέη που είναι υπεύθυνο για, το... για την πολιτική αλληλεία στο, Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο γιατί πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές και από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκαν σε θέματα που θα ήθελα να θίξω και εγώ. Ε, νομίζω ότι πρέπει πρώτα πρώτα να πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χαιρετίζει το γεγονός ότι τόσο νωρίς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α, αρχίζει η συζήτηση για τις μελλοντικέ αλλαγές. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι στις συζητήσεις αυτές θα ακουστούν και οι γνώμες άλλων κρατών μελών και αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπέρ μιας πολιτικής, μια, ε, ε είναι υπέρ της μεταρρύθμισης της κοινής πολιτικής αλίας. Ε, δεν ε, είναι ότι Ε, δεν είναι ότι λέμε ότι όλα πάνε στραβά όπως είπε ο κύριος Μπόργκ αντιθέτως η διαχείριση είναι πολύ δύσκολη, περίπλοκη και είναι γεγονός ότι η πολιτική ε, αυτή είναι κοινή ασχολούμεθα με κοινού ε, πόρους και πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ε, για το πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που είδαμε ότι υπάρχουν παραδείγματος χάρη απορρίψεις ε, ε, μη δηλω θέντα αλλιεύματα ανεξέλεγκτα κλπ. Ε, εμείς λέμε ότι η κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητική γι' αυτό συμφωνούμε με τα συμπεράσματα των ε, Υπουργών του περασμένου Σεπτεμβρίου ε, την ανάγκη για μεταρρύθμιση και εν πολύ στα αποτελέσματα της ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν χρειάζεται να επαναλάβω πολλά από τα σημεία με τα για τα οποία συμφωνούμε με τον Επίτροπο Μπόρκ. Είναι προφανές ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι, δεν θα λυθούν όλα με τη μεταρρύθμιση αλλά πολλά μπορούν να ξεπεραστούν χρειαζόμαστε ίσως καινούριε κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να ε, ορίσουμε τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές Πιστεύουμε ότι οι πολλά ε, μπορούν να αποφασίζονται και να εκτελούνται σε διαφορετικά επίπεδα. Θέλουμε η δίκαιη και ε, αναλογική ε, πρόσβαση σε πόρους και αποθέματα και προσπαθούμε για μια για ένα βιώσιμο κλάδο. Ε, εμείς οι περισσότεροι μάλλον από μας που ασχολούνται με πολιτική ε, ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα και πώς θα επιτευθούν αυτά και όχι για τα εργαλεία με τα οποία θα επιτευθούν οι στόχοι. Γι' αυτό χάρηκα που ο κύριος Μπόρκμα έδωσε, είπε ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες εξουσίες, δικαιοδοσίες και ευθύνες ε, στον ίδιο τον κλάδο της αλίας. Μιλάμε για μια πολιτική η οποία πέραν της ε, των οικονομικών στόχων έχει και στόχους που σχετίζονται με τη διατήρηση των αποθεμάτων και την και την ε, ε, βιωσιμότητα του και την προστασία του περιβάλλοντος με πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να καλυφθούν και γι' αυτό οι στόχοι θα πρέπει να είναι περισσότεροι από αυτούς που είχαμε μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ καλό που θα γίνει συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα ο Χιούρανκεν Ντέιβις, ο υπουργό μας στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα ε, είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελε να παίξει ένα ε, σημαντικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής αλίας. Αντί να έχουμε ετήσιες διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουμε περισσότερες επαφές, περισσότερες διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Ο κλάδος θα πρέπει να αναλάβει ε, περισσότερες ευθύνες και η η πολιτική θα πρέπει να ε, ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιφερειών ούτω ώστε να μπορούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη να έχουμε μια πολιτική η οποία θα, παρα, θα οδηγήσει, θα δώσει τους καρπούς που επιθυμούμε όλοι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο να φτάσουμε το όραμα αυτό Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε 10 λεπτά για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Αν δεν έχετε κάποια ερώτηση και απάντηση προς αυτή την ενότητα, α, δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση για τον Χιούγκο Άντερσον. Όσον αφορά τα γνωμοδοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, είπε ότι έχουν τέτοια δομή αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να του αναθέσουμε και διαχείριση. Και ε, παρέθεσε τις ε, ε, περιφερειακές μονάδες διαχείρισης στις Ηνωμένε Πολιτείε. Τι πιστεύετε. Σε νέες μονάδες διαχείρισης τι βαθμό διαχείρισης μπορούμε να αναθέσουμε. Μιλώ για νέες μονάδες, ε, όπως το, ε, ακολουθώντας το παράδειγμα τον είπα. Πιστεύετε ότι η συνολική διαχείριση θα μπορούσε να αναλυφθεί από αυτούς τους περιφερειακούς φορείς, ενώ η Επιτροπή στα πλαίσια της συνθήκης θα ε, παραμείνει ως διαιτητής, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η ισοτιμία στην οποία αναφέρθηκαν οι ομιλητές. Γιατί αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αυτό το κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης. Κύριε Άτγουλ, ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Άντερσον και εγώ. Πολύ παρόμοια με την ερώτηση του κύριου Στίβενσον μιλήσατε για τα περιφερειακά γνωμοτικά συμβούλια, τα οποία με την παρουσία του μορφή δεν, θα είναι σε θέση να αναλάβουν βασικέ ευθύνε, αρμοδιότητε διαχείριση. Συμφωνώ απόλυτα. Ιδιαίτερα ω προ τη χρηματοδότηση. Και ελπίζω να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Αλλά, κοιτάξτε, αν θέλουμε να αναθέσουμε τη διαχείριση σε κάποιου φορεί διαχείριση, ποιο θα είναι ο ρόλο των περιφερειακών γνωμοτικών συμβουλίων. και πού θα λαμβάνω δύο αποφάσει περί διαχείριση. Και έχω και μια ερώτηση προ τον κύριο Σου. Είπατε ότι ω προ τα ITQ, Τι επιμέρους ποσοστώσεις, ατομικές ποσοστώσεις, ε, εδώ ε, πρέπει να το δούμε το θέμα, ε, πρέπει να δούμε χωριστά το θέμα για τα πελαγικά είδη έναντι των λευκών ψαριών. Γιατί ε, ε, ε, πώς το βλέπετε, το βλέπετε σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των λευκών ψαριών που είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο ελίας. Η κυρία Φράγκα. Και εγώ θέλω να μιλήσω με το περίφημο θέμα της αύξησης των αρμοδιοτήτων των ΡΑΚ, των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων. Εγώ, όπως και ο κύριος Άντερσον, πιστεύω ότι λαμβάνοντα υπόψη τι αρμοδιότητε τι υφιστάμενε αρμοδιότητε των γνωμοδοτικών ε, συμβουλίων, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να του αυξήσουμε τι αρμοδιότητε. Αλλά είναι αλήθεια ότι στην μεταρρύθμιση, και εγώ θέλω να συζητήσω το θέμα, τουλάχιστον όταν θα φτάσουμε στη μεταρρύθμιση. Ε, αναφέρεται πιθανότητα αλλαγή των αρμοδιοτήτων σε διάφορα επίπεδα. Τώρα, θέτουμε το ερώτημα των αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμών, των κρατών μελών, και των αρμοδιοτήτων που θα μπορούσαν να εκχωρηθούν σε περιφερειακό επίπεδο και μια άλλη κατανομή ενδεχομένω. Ρωτώ, για να αυξήσουμε τι αρμοδιότητε σε περιφερειακό επίπεδο, τότε θα πρέπει να αφαιρέσουμε αρμοδιότητε από τα κράτη-μέλη, έτσι δεν είναι. Θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη ή όχι. Ρωτώ, επειδή εδώ έχουμε εκπροσώπου των κρατών μελών. Ποια είναι η άποψή του. Γιατί το να δώσουμε περισσότερε αρμοδιότητε σε, σε κάποιου σημαίνει αφαίρεση αρμοδιότητε από κάποιου αρμοδιοτήτων από κάποιου άλλου. Και θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Γιατί το είπε πολύ καλά ο κύριος Άντερσον. Έχουμε ένα μοντέλο στη ΣΥΠΑ που είναι τελείως διαφορετικό από το δικό μας. Οι περιφερειακέ επιτροπέ των ε, ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά ΡΑΚ, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Και όλα αυτά συνδέονται με το συνολικό πρόβλημα έλλειψη ε, διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Μα είπε ο πρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είναι υπέρ τη βιωσιμότητα ε, και θέλει να δούμε αυτή τη μέγιστη διαρκή απόδοση. Αλλά κοιτάξτε, ε, οι υπουργοί μιλούν για τάκ και για ποσοστώσει και πολύ συχνά παίρνουν αποφάσει που έρχονται σε αντίθεση με τι μέγιστε διαρκεί αποδόσει και με τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Πολύ ωραία. Ε, να δώσουμε το λόγο στου τρει εμπειρογνώμονε. Σα υπενθυμίζω. Δέκα λεπτά για τι απαντήσει. Αλλά ήδη έχουν περάσει τα 3,5 λεπτά από αυτά τα 10. Κύριο Άντερσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όπως είπε και ο κύριος Στίβενσον, είναι το βασικό ερώτημα. Η οργάνωση δηλαδή και η δομή. Αλλά όπως βλέπω εγώ το θέμα, η βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τη συνολική πολιτική που δηλώνει τις βάσεις της πολιτικής δομέας της Αλίας. Στα επόμενα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό, όλα αυτά τα επίπεδα, τηρούνται αυτές οι δεσμεύσεις και γίνεται διαχείριση. Να αναφερθώ και πάλι στο παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την οδό ακολουθούν. Υπάρχει δηλαδή μια ομοσπονδιακή συνολική πολιτική και μετά η διαχείριση γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Η διαφορά είναι ότι τα περιφερειακά αυτά όργανα εκλέγονται και εκπροσωπούν ε, πολλούς ενδιαφερόμενους, όπως και εμείς τα ΡΑΞ, αλλά έχουν τους δικούς τους πόρους κτλ. Έχουν τους πόρους δηλαδή για την αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων τους. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των νομοθετικών συμβουλίων. Όσον αφορά τη δομή τους, είναι θελοντικές. Δηλαδή, αν κάποιες ε, στη δική μας την περίπτωση είναι θελοντική η συμμετοχή. Ε, οι, οργανώσεις αποφασίζουν ότι ε, θέλουν να είναι και μέλη του ΡΑΚ, του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Το μελλοντικό τους ρόλο. Τα ΡΑΚ φυσικά ε, θα εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο των γνωμοδοτικών συμβουλίων. Ενδεχομένως, εκτός από το ότι μπορεί και να είναι διαχειριστικά, ε, διαχειριστικά όργανα σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί όπως είπε η κυρία Φράγκα, δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα δεχτούν να μην εμπλέκονται σε περιφερειακό επίπεδο. και να αφήσουν ολοκληρωτικά τη διαχείριση της ελευθερικής πολιτικής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και στη βιομηχανία. δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Άρα μάλλον θα πρέπει να συμμετάσχουν και τα κράτη-μέλη ναι. σε περιφερειακό επίπεδο. Ίσως όμως ο κύριος Σου μπορεί να το σχολιάσει. Γιατί εκπροσωπεί την κυβέρνηση της Δανίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η, η αλληλεία των πελαγικών ναι είναι πολύ σημαντική. Αν λάβουμε υπόψη ε, ότι πρόκειται για είδη ε, που έχουν χαμηλές τιμές και είναι μεγάλα σε αριθμό. Ε, η πολιτική μας είναι ότι όσον αφορά τα ITQ στα πελαγικά πρέπει να έχουμε ένα σαφέστατο, ξεκάθαρο σύστημα. Η πολιτική της Δανίας λοιπόν είναι τέτοια που θέλουμε να έχουμε παράκτη αλία, θέλουμε να υποστηρίξουμε τους νεοαφιχθέντες στον κλάδο και θέλουμε ποικιλία ε, στο στόλο. Πριμοδοτούμε λοιπόν την παράκτη αλία και τους νέους που ασχολούνται με την αλία. Αυτή η πολιτική έχει δώσει, έχει δώσει αποτελέσματα. Ο λόγος τον οποίο οδήγησε συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι γιατί όταν η αλληλεία ε, είναι αποδοτική, τότε εξοικονομούνται χρήματα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε τι προτεραιότητέ μα. Ναι. Το, ε, Υπουργείο, το, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών τη Δανία υπολόγισε ότι περνώντα από το παλιό σύστημα διαχείριση το σύστημα ITQ, απελευθερώνται κάθε χρόνο 60 εκατομμύρια ε, ευρώ. τα οποία τα ε, γιατί εξοικονομούνται από, από πλοία τα οποία πλέον δεν αλλιεύουν ανώφελα και καύσιμο το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Τα χρήματα αυτά λοιπόν πηγαίνουν σε άλλους σκοπούς. Είναι λοιπόν συγκεκριμένη επιλογή πολιτικής. Πολιτική επιλογή μάλλον. Όσον αφορά τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, να σας πω ότι κατά την άποψη της κυβέρνησης της χώρας μου, τα συμβούλια αυτά παίζουν ουσιαστικό ρόλο ως προς την ε, ε, ε, εφαρμογή των στρατηγικών και κατευθυντηρίων γραμμών της κοινή ελληνικής πολιτικής. Αλλά όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση σε επίπεδο αλλιέως, αυτά πρέπει να αφήσουμε στους επιμέρους αλλιείς, σύμφωνα με αυτά που σας είπα και προηγουμένως. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη ενότητα. Κύριος Γκεράν, Γενικός Γραμματέας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού ε, Συμβουλίου για τα Δυτικά Ήδατα του Νότου. Ο κύριος Λεσνέ από το ε, Υπουργείο Γεωργίας και Αλίας της Γαλλίας και ο κύριος Μοντέιρο, Γενικός Διευθυντής ε, Αλίας Ιδατοκαλλιέργειας από το Υπουργείο Γεωργίας ε, Ανάπτυξη Πέθρου και Αλίας Πορτογαλίας. Κύριος Γκέραν για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Αλίας του Κοινοβουλίου που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα. Όπως και ο Ούγκο Άντερσον δεν θα σας ε, παρουσιάσω τη λεπτομερή θέση μας για την αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής γιατί αναμένουμε ακόμη την πράσινη βίβλο αλλά θα βασιστώ σε γνωματοτήσεις που έχουν ήδη δοθεί από την οργάνωσή μου. Το ΣΕΣΕΑΡΣΟΥ είναι μια δομή που δημιουργήθηκε πολύ πρόσφατα τον Απρίλιο 2007 αλλά προϋπήρχε πριν από ένα χρόνο είχαν ακούσει οι πρώτες ιδέες. Προέρχεται από την προηγούμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΛ που είχε σαν στόχο την προσέγγιση των διαφόρων αλλιευτικών πολιτικών. Είχε μόνο συμβουλευτικό ρόλο τότε. Είναι καταρχήν γεωγραφική η προσέγγιση του διότι βασιζόταν στην διαχείριση, κοινή διαχείριση των ελληνικών πόρων ή των αποθεμάτων για να συνομιλούν εκεί ελεύθερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον ίδιο πόρο, δηλαδή τους ηχθείες. Όλοι γνωρίζουν τη σύνθεση του Συμβουλίου αυτού κατά ένα τρίτο οι ενδιαφερόμενοι και κατά τα δύο τρίτα οι επίσημοι. Και είναι τελείως θελοντική η συμμετοχή. Τώρα ορισμένα θετικά στοιχεία για τη λειτουργία του μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας. Καταρχήν η αντιπροσωπευτικότητα. 106 οργανώσεις είναι μέλη του. Αν και ακόμη λείπουν ορισμένες από το Κάντιθ, από τα Σκαναρίους, ή από τη μεταποιητική βιομηχανία. Υπάρχει διάθεση των πληροφοριών σε όλους όσους ενδιαφέρονται και που μπορούν έτσι να έχουν μια κοινή κατανόηση και ανάλυση των μηχανισμών που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι όπως ξέρουμε δεν κατανοούν όλοι με τον ίδιο τρόπο τα ίδια πράγματα. Και τέλος αποτελεί ένα βήμα ανταλλαγή απόψεων που δεν έχει προηγούμενο και επιτρέπει ένα διάλογο παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν γιατί έχουμε τέσσερις γλώσσες εργασίας, τεράστιος αριθμός. Τώρα, η συμμετοχή των μίκη ομικρόν. Πολύ συχνά οι επαγγελματίες ζητούν από το ΣΕΣΕΡ να διοργανώσει συζητήσεις για κάποιο πρόβλημα και φυσικά εμείς με τη σειρά μας ζητούμε γνωμοδότηση από τη ΜΚΟ όμικρον για να φέρουμε εκεί μαζί όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συνεργασία των χωρών μελών και των επιστημόνων, εμείς είμαστε πολύ καινούργια οργάνωση βέβαια και η συνεργασία αυτή αρχίζει μόλις να δημιουργείται Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά, αλλά διαπιστώνουμε ήδη ότι όλο και περισσότερες οργανώσεις συνεδριάζουν για να συζητήσουν το ίδιο θέμα. Υπάρχει επικάλυψη δηλαδή τέλος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κατάλληλους Κομισιών. Ε, ο κύριος στόχος μας βέβαια είναι να δούμε αν θα έχουν λόγο τελικά στα μάτια της Κομισιόν. Εδώ και πολλούς μήνες βλέπω ότι μειώνεται ο ενθουσιασμός των μελών και υπάρχει ο κίνδυνος να μπούμε σε έναν φαύλο κύκλο όπου οι απαντήσεις της Κομισιόν που πολλές φορές είναι τελείως άσχετες από τα ερωτήματα που τίθενται θα δημιουργήσουν ακόμη λιγότερο ενθουσιασμό. Πολλές φορές οι απαντήσεις αυτές είναι απλώς ευγενείς απαντήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα. Έτσι λοιπόν το ένα θα φέρνει το άλλο και αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν αμοιβέ, να ικανοποιούνται αμοιβέ ανάγκες. Συμβατέ βέβαια με την κάλπα, αλλά και οι απαντήσεις τη Κομισιόν να σέβονται ένα, κάποια ορισμένη διοντολογία. Για να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο προτείνουμε κάτι σωστότερο. Έναν μη φαύλο κύκλο δηλαδή. Τα τρία μέρη, δηλαδή η λήψη αποφάσεων με τις διοικήσεις και την Κομισιόν, οι επιστήμονες και οι αλληλείς, να συνεννοούνται καλύτερα. Καταρχήν σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο, γιατί επί της ουσίας η συνεργασία αυτή θα επέτρεπε την ανταλλαγή ε, απόψεων που να καταλήγουν σε αποφάσεις με κύριο στόχο βέβαια μια έγκριση από, με μορφή κανονισμού από την Ένωση και συμβολικά η υπογραφή συμφωνίας διαχείρισης μακροπρόθεσμα μεταξύ και των τριών πλευρών θα έδινε πολύ μεγαλύτερη ορατότητα και εμπιστοσύνη και στα τρία μέρη, συμβαλόμενα μέρη και θα μπορούσαν όλοι να είναι βέβαιοι ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει ατομικές και συλλογικές δεν θα έχουν πάει χαμένες και θα καταλήξουν σε σύνταξη συγκεκριμένων προοπτικών. Για τα σχέδια διαχείρισης ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα Έχουμε γράψει μία μπροσούρα που τη στείλαμε και σε πολλούς κοινοβουλευτικούς των χωρών μελών που συμμετέχουν και το θέμα είναι σε ποια κλίμακα θα εργαστούμε. Σε κλίμακα κάποιας συγκεκριμένης αλλιευτικής κοινότητας αλλά να συμμετάσχουν σε αυτό όλοι. Άρα να υπάρχει και κάποια διοικητικό συμβούλιο και ένα συντονιστή που δεν υπάρχει ακόμη και που να είναι σε θέση να παρακολουθεί όλες τις φάσεις της νομοθετικής διαδικασίας όσο δύσκολη και να είναι η κατανόησή τους και τέλος την εμπειρική γνώση που έχει ο τομέας να την διατυπώσει πιο επίσημα έτσι ώστε οι στόχοι που είναι και οικολογικοί και οικονομικοί και κοινωνικοί να συνδυαστούν με κύρια ιδέα να υπάρξει ένα συλλογικό πρόγραμμα αλλά με κάποια ελαστικότητα γιατί οι πόροι που μας ενδιαφέρουν, οι ηχθείες δηλαδή είναι κάτι που διακυμαίνεται και να υπάρχει σαφής διατύπωση του κοινού στόχου. Νομίζω ότι ένας, μια τέτοια οργάνωση θα μπορούσε να επιτρέψει περισσότερη προβλεψιμότητα και συνεννόηση για να βγούμε από, τις, από τα απρόβλεπτα στοιχεία που πλήττουν συνέχεια την ΚΑΟΠ. Και τέλος να παρακολουθεί και το πώς εφαρμόζονται οι κανονισμοί αφού θα παρακολουθεί στενά όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τώρα ορισμένες λέξεις κλειδιά όλα τα συμβαλώμενα μέρη αλλά και οι διοικήσεις και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν επιστήμονες άλλο η υπευθυνότητα ή ο σχεδιασμός και κατά τα άλλα για το ΣΕΣΕΡΣΟΥΝΤ θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα Interreg για να συνδέσουμε και το ΣΕΣΕΡ και τους επιστήμονες και τις εθνικές διοικήσεις και το πρόγραμμα, το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί από το 10 μέχρι το 12. Δηλαδή μέχρι την κατάληξη της πρώτης φάσης της μεταρρύθμισης. Έχουμε βέβαια τα υπόλοιπα στην ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκέρα. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λενέ που είναι ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αλίας και Ιρδοκαλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας και Αλίας της Γαλλίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για το γεγονός ότι προσκαλέσατε τη Γαλλία να τοποθετεί στη σημερινή ακρόαση. Όπως αναφέρετε κι εσείς, έλαβαν χώρα οι πρώτες ανταλλαγές απόψεων επί Γαλλικής Προεδρίας έχουμε, ε, τώρα ξεκινάμε ένα νέο στάδιο, της, αυτό της δημόσιας διαβούλευσης μετά από την ανταλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Ευχαριστούμε λοιπόν την Επιτροπή ε, για την μελλοντική παρουσίαση της Πράσινης Βίβλου που θα αποτελέσει τη βάση ε, ε, χρήσιμων ανταλλαγών. Το περασμένο Σεπτέμβριο οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και έτσι μας δόθηκε ευκαιρία να προβληματιστούμε σε ορισμένα βασικά ζητήματα. η επιστημονική διάσκεψη για τους αλληλείς που οργανώθηκε στο Κοινοβούλιο επέτρεψε επίσης ε, να ε, ανταλλαγούν απόψεις για ορισμένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βαθύνουμε περαιτέρω. Όσον αφορά πρώτα απ' όλα τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί η Γαλλία, κυρίως ε, όσον αφορά την κατάσταση των αποθεμάτων ή το ζήτημα της υπεραλίευσης. Οι βασικές αιτίες αυτής της κατάστασης εντοπίζονται την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας βρίσκουν σύμφωνους οι διαπιστώσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάπως ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε ότι ε, καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες από τα κράτη-μέλη ε, από το διάστημα που μεσολάβησε από τη μεταρρύθμιση του 2002. Βεβαίως η κατάσταση των αποθεμάτων σαφώς και δεν μας ικανοποιεί, το αντίθετο. Ορισμένα αποθέματα βρίσκονται εκτός των ε, βιολογικών ορίων ασφαλείας, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ε, έχει αντιστραφεί η πτωτική τάση που ακολουθούσε η βιομάζα και έχει ξεκινήσει η μείωση της ελληνικής ικανότητας σε πολλές περιπτώσεις. Βεβαίως τα αποτελέσματα δεν, τα, ε, δεν μπορούν να γίνουν αισθητά, αλλά ε, είναι σίγουρο ότι θα, όλα αυτά θα επιδράσουν με θετικό τρόπο. Η βελτίωση αυτή των αποτελεσμάτων δεν έγινε τυχαία. Η Γαλλία και πολλά άλλα κράτη-μέλη κατέβαλαν πολύ σημαντικέ οικονομικέ προσπάθειε για να αναπτύξουν συγκεκριμένα προγράμματα ε, μείωση τη ε, υπεραλίευση ορισμένων ε, αλλιευτικών στόλων. Όλα αυτά εντάσσονται στα πλαίσια μια γενικότερη λογική ρύθμισης τη πρόσβαση μέσω της, ε, ε, θέσπιση συγκεκριμένων συστημάτων και αδειών για να μην ξαναγυρίσουμε στην κατάσταση της υπεραλίευσης. Ε, στα, ε, στις περιπτώσεις ε, που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά. Γενικότερα, διαπιστώνω ότι τονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αρνητικός ρόλος των επιδόσεων στον κλάδο αυτό. Αλλά αυτή η διαπίστωση είναι υπερβολικά γενική. Τα, τα, τα, τα δημόσια κονδύλια θα μπορούσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να προσανατολίζονται σωστά οι επενδύσεις. Ακριβώς αυτό υπάρχει το Ταμείο για την Αλία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ισχυρό κινητήριο μοχλό για να διοχετευτούν οι επενδύσει και οι έρευνε προ την κατεύθυνση επίτευξη καλών αποτελεσμάτων. Με τη μεταρρύθμιση του 2002 ε, ε, ε, ετέθησαν οι τελείω διαφορετικέ οικονομικέ συνθήκε για τι επιχειρήσει και οι συνέπειε μόνο μεσοπρόθεσμα θα δείξουν τα, θα, δείξουν, τα αποτελέσματά του. Να πω τώρα το εξή όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των ηλεκτρικών πόρων. Αυτό είναι κοινό στόχο. Όμω, ε, ακούγοντα ορισμένε τοποθετήσει για το θέμα τη αλληλεία, αναρωτιέμαι για το κατά πόσον υπάρχει η βούληση ε, διατήρηση του τομέα τη αλεία, συγγνώμη. Απέναντι στο ερώτημα αυτό, η Γαλλία θέλει να απαντήσει χωρί υπεκφυγέ. Η αλληλεία ε, ε, οδηγεί ε, στην παροχή τροφίμων ποιοτικών και ποσοτικών. Και δεν μπορούμε ε, και δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε και να υποκαταστήσουμε την αλεία. Αυτά μπορεί να σα φαίνονται στοιχειώδη, αλλά έχουν συγκεκριμένε συνέπειε. Οι περιβαλλοντολογικέ επιπτώσει θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ελεγχθούν, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα ε, και να γίνουν αποδεκτέ να γίνουν αποδεκτέ η κοινωνική διάσταση και η οικονομική διάσταση, γιατί δεν μπορούμε να τι παραμελήσουμε τι συνιστώσει αυτέ στα πλαίσια τη ανάλυση μα. Τώρα, να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία τα οποία πιστεύω ότι είναι θεμελιώδη όσον αφορά την πρόσβαση στα ύδατα και στους πόρους. Για την γεωγραφική πρόσβαση. Το καθεστώς των 6 και 12 μιλίων σήμερα δεν αμφισβητείται στο μέτρο που προέρχεται από μια ισορροπία που επιτρέπει τη διατήρηση του βιοτεχνικού παράκτιου στόλου Άρα λοιπόν στις παράκτιες ζώνες θα μπορούν να δρουν οι επαγγελματίες που είναι σε τελευταία ανάλυση οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Όσον αφορά την πρόσβαση στους πόρους, το θέμα αυτό συνδυάζεται και σχετίζεται άμεσα με τις λεπτομέρειες ε, ε, διαχείρισης. Τα μέτρα διαχείριση, όπω υπογράμμισε η κύρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περνούν από ανάληψη ευθύνη από του ίδιου επαγγελματίε. Αυτά τα μέτρα λοιπόν πρέπει να λάβουν υπόψη την μεγάλη ποικιλομορφία των αλλιευτικών στόλων και τον ε, ε, ποικίλο χαρακτήρα τους, αλλά και και βεβαίως ε, εδώ θα πρέπει να βρούμε μεθόδους που να προσαρμόζονται στις επιμέρους πραγματικότητες των επαγγελματιών ε, και να οδηγούν σε ισότιμη αντιμετώπιση, εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς τρέβλωση της αγοράς και χωρίς να ε, επανερχόμαστε στην αρχή της ε, σχετικής σταθερότητας στην οποία στηρίζεται η κοινή πολιτική ελίας. Τώρα, όσον αφορά ε, ε τις εξελίξεις του συστήματος που είναι απαραίτητες, αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν στην, στην, στο συντονισμό της διαχείρισης με τις ελευτικές προσπάθειες. Οι κανόνες διαχείρισης θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε ε, να έχουμε μία μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση και, ε, ε, και η πολιτική αυτή να μην αποτελεί αντικείμενο αναθεώρηση κάθε χρόνο, η πολιτική διαχείριση. Αντίθετα, λαμβάνοντα υπόψη ε, τη διακύμανση των περιβαλλοντολογικών όρων, θα πρέπει τα όρια και τα επίπεδα να ορίζονται τήσια. Η κοινή πολιτική στο τομέα τη Αλία θα στεφτεί από επιτυχία μόνο εάν η διάγνωση των οικοσυστημάτων και των, και των αποθεμάτων είναι κοινή. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χώρο ανταλλαγή απόψεων και να ενισχυθεί η εταιρική σχέση μεταξύ των επιστημόνων και των αλλιέων σε κοινοτικό επίπεδο. Να προωθήσουμε ε, τη δυναμική συνεργασία των δύο αυτών πλευρών. Να ενθαρρύνουμε τους επαγγελματίες οι οποίοι θα πρέπει να βοηθήσουν την έρευνα συλλέγοντας στοιχεία. Από την πλευρά τους οι ερευνητές θα πρέπει να, ενθαρρύνουν, να ενθαρρύνονται έτσι ώστε να στρέφονται προς ίδιους επαγγελματίες. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των παραμέτρων όπως, ε, ε, ε, όπως προκύπτουν κατά την επεξεργασία της νομοθεσίας. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στους βιολογικού παράγοντες, περιβαλλοντολογικού, οικονομικού και κοινωνικούς. Η, η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων και η βελτίωση του διαλόγου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας τέτοιας δημόσιας πολιτικής. Και η σημερινή άλλωστε ακρόαση συμβάλλει στο στόχο αυτό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ευρεία διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση τη κοινή πολιτική στον τομέα τη Αλία. Η μεταρρύθμιση του 2002 δημιούργησε ε, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, τα οποία αποτελούν πλατφόρμα συζήτηση, προβληματισμού και ανάλυση. Τα θεσμικά πλαίσια ε, πρέπει όμως να τροποποιηθούν κυρίω με το πέρασμα ε, τη συναπόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα καλεί να μελετήσουμε διάφορε δυνατότητε επίπεδο λήψη απόφαση. Από το σημερινό επίπεδο ε, λήψη αποφάσεων στου υπουργού ε, μέσω τη ανάληψη ευθυνών από όλου του εμπλεκόμενου μέσω τη διαδικασία επιτροπολογία. Θα πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε όλε αυτέ τι δυνατότητε. Θα πρέπει όμω να τονίσουμε ότι η συνέπεια των κοινοτικών πολιτικών δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσω τη διατήρηση του βασικού ρόλου που είναι υπεύθυνα, του βασικού ρόλου των κρατών μελών που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και τον έλεγχο των πολιτικών. Υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε τι διάφορε αναλυτικέ λύσει. Η συζήτηση για τον κανονισμό για τους ελέγχους και τα τεχνικά μέτρα τα οποία υπάρχουν σήμερα θα μας επιτρέψουν μέχρι να γίνει η επόμενη αναθεώρηση να φτάσουμε σε συνένεση. Πάντως απαιτείται απλοποίηση καθώς επίσης και λήψη υπόψη ε, των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της Ελίας. Τίθεται όμως το εξής ερώτημα όσον αφορά ε, τη, τη συσχέτιση αυτής της ε, μεταρρύθμισης με, την, με, το, με το μέλλον της κοινή πολιτικής στον τομέα της Ελίας. Σήμερα έχουμε βαθιές αλλαγές. Οι ενεργειακές προκλήσεις, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Απέναντι στα προβλήματα αυτά γιατί να εγκαταλείψουμε οποιαδήποτε ιδέα δημόσια παρέμβαση στον τομέα τη αλεία. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι απαιτείται ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στον τομέα τη αλεία, συνεπή με τι βασικέ αρχέ τη ε, διατήρηση των ειδών, που να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ε, ε, παγίωση τη διαρκού αλεία. Όσον αφορά τι διεθνεί σχέσει, να υπενθυμίσω το βασικό ρόλο που έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει η ευρωπαϊκή κοινότητα στη διεθνή σκηνή στα πλαίσια των διμερών σχέσεων, αλλά και διαμέσου της συμμετοχής της στα πολυμερή φόρα. Ε, η κοινότητα συμβάλλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο. Εν συμπεράσματι θα ήθελα να υπογραμμίσω τα σημεία κλειδιά ε, για την επιτυχία ε, της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Εντοπισμός σαφών και συγκεκριμένων στόχων ε, ε, λήψη αποφάσεων στο επαρκέ επίπεδο, έτσι ώστε ε, να υπάρχει απαραίτητη προσαρμογή με όλε τι συνδεδεμένε πολιτικέ, σύνδεση τη έρευνα με του επαγγελματίε, να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερότητε των διαφόρων τομέων αλίας και ιδιαίτερα τη ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στις ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιφέρειες, ενθάρρυνση για την προσαρμογή των στόλων στις οικονομικές πραγματικότητε και στι περιβαλλοντικέ ανησυχίε. Αυτά και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ουρίκο Μοντέιρο που είναι Γενικός Διευθυντής Αλληλείας και Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας και Αρχής της Υπέθρου της Πορτογαλίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την Επιτροπή Αλίας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε. Είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της κοινότητας. Η μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής ε, είναι ε, σημείο κλειδί για το μέλλον της ε, κοινότητας και βεβαίως στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει μια θέση ε, για το θέμα αυτό επανειλημμένος. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ε, ποια είναι η κοινή αυτή πολιτική, τι επετεύχθη το μεταξύ και τι όχι μετά τη μεταρρύθμιση του 2002. Τώρα μιλάμε για μια καινούργια μεταρρύθμιση το 2012 η οποία έχει σαν στόχο να επιτύχει πραγματικά μια βιώσιμη ε, αλία. Η τωρινή κοινή πολιτική αλίας πραγματικά έχει ξεπεραστεί παρόλο που έγιναν σημαντικές πρόοδοι και όλος η διαχείριση των ε, αποθεμάτων ε, σε πολυετή βάση, η δημιουργία των γνωμοδοτικών, περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων. Όλα αυτά είναι θετικά πράγματα τα οποία πέτυχε η πολιτική αλίας που ισχύει αυτή τη στιγμή. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να δούμε από εδώ και μπρος είναι οι άλλοι τομείς όπου δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο θετικοί ο αλευτικός τόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, είπαν και προηγούμενοι ομιλητές η κατάσταση των αποθεμάτων η κατάσταση των αλληλευτικών πόρων αυτά είναι πράγματα που μας ανησυχούν και ξέρουμε ότι γίνεται υπεραλίευση ε, τουλάχιστον για ορισμένα είδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε το σωστό τρόπο και τον πιο γρήγορο τρόπο τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε 7 ε, θέματα τα οποία είναι κατά την άποψή μου σημαντικά και βεβαίως θα μπορούσα να απαντήσω και για άλλα θέματα αν υπάρχουν ερωτήσεις. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι η διαχείριση των αποθεμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ισορροπία θέλουμε να επιτύχουμε και με ποιο τρόπο η, τα μέγιστα, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα, τα τάκ και δηλαδή που εφαρμόζονταν μέχρι τώρα μπορεί να δούλευαν στο παρελθόν αλλά αυτό τι τη στιγμή έχουν ξεπεραστεί. Δεν είναι δυνατόν με βάση τα τάξη και τα κουότας να προχωρήσουμε στη διαχείριση ένα είδος παραδείγματος χάρη. Η... Επειδή εντωμεταξύ δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει την ε, δραστηριο... 100% δραστηριότητα του αλλιευτικού στόλου ε, γι' αυτό τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο εμείς πιστεύουμε ότι η οργάνωση της αλλιευτικής προσπάθειας με το σωστό τρόπο, με τα σωστά εργαλεία, με τη σωστή τεχνολογία με λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτερότητες ορισμένων περιοχών ε, είναι καλύτερος τρόπος ε, να προχωρήσουμε από ότι τα τάξ και οι ποσοστώσεις. Βεβαίω αυτό δεν ε, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επιθεωρήσεις, έλεγχη και παρακολούθηση των επιστημονικών στοιχείων. Δεύτερο θέμα είναι η, που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η προσαρμογή της δυναμικότητας ανάλογα με την περιοχή και με το είδος. Ξέρουμε ότι η θνησιμότητα των ε, ειδών διαφέρει και, αλλά είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη αν θέλουμε να προχωρήσουμε θετικά η Πορτογαλία αυτό το λαμβάνει υπόψη και προσπαθεί γι' αυτό να προσαρμόσει τη δυναμικότητα του στόλου της ε, από το 2004 και μετά ε, ε ξέρουμε ότι δεν δίνονται πλέον ενισχύσεις για την κατασκευή νέων αλλιευτικών σκαφών συγκεκριμένου είδους και ε, ε, είδαμε πόσο μειώθηκε ο πώς εξελίχθηκε ο στόλος της ε, κοινότητας με το με τον αφοπλισμό των παλαιών σκαφών που τελικά έπρεπε να εξυγχρονιστούν ε, τα, τα οποία είτε παροπλίστηκαν τελείως είτε αντικαταστάθηκαν από πιο σύγχρονα. βεβαίως ε, εκεί υπάρχει και οικονομικό πρόβλημα για τους ε, ιδιοκτήτες των σκαφών το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ωστόσο πιστεύουμε ότι στόχος μας πρέπει να είναι ένας πιο σύγχρονος και πιο ευέλικτος αλλιευτικός στόλος. Βεβαίως εδώ δεν υπάρχουν λύσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα ε, Υπάρχουν α, όμως κάποιες απαρχές λύσεις που έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Επόμενο θέμα, η πρόσβαση, ίση πρόσβαση και ελεύθερη πρόσβαση σε ύδατα και πόρους. Η, αυτή είναι μια βασική αρχή της κοινή πολιτικής αλίας υπάρχουν επίσης υπάρχει η αρχή των 12 μιλίων για την ε, αλλιευτική έκτημα που εφαρμόζει στις ορισμένες ε, περιοχές οι οποίες ε, οποία είναι σεβαστή και χρήσιμη Αυτές οι αρχές λοιπόν πρέπει να διατηρηθούν. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα της υπεραλίευσης άρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα συγχρόνως ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν από την αλία η οποία ήταν, είναι στις περιοχές αυτές παραδοσιακή δραστηριότητα εδώ πρέπει να προσέξουμε το επόμενο θέμα είναι το θέμα της σχετικής σταθερότητας που είναι άλλη βασική αρχή της κοινή πολιτικής αλίας βεβαίως χρειάζεται ε, να διατηρηθεί η αρχή αυτή και συγχρόνως πρέπει να επαγρυπνούμε και σχετικά με τη διατήρηση κάποιων δικαιωμάτων, του σεβασμό κάποιων δικαιωμάτων ναι. κρατών μελών. Στα διάφορα κράτη-μέλη τα πράγματα είναι διαφορετικά και εδώ χρειάζεται λοιπόν μια ευέλικτη προσέγγιση διότι οι λύσεις που θα μπορούσαν να επιτύχουν στο α κράτος μέλος ίσως αποτύχουν στο β. Ε, για το θέμα της εμπορευσιμότητας κάποιων δικαιωμάτων το οποίο φαίνεται να συζητείται αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία έχει πάρει θέση λέμε ότι Κύριε Μοντέιρο πιστεύω ότι επειδή τώρα έχουμε 10 λεπτά για να απαντήσουμε ε, τότε ε, εάν σας έμεινε κάτι, ε, στα, ε, το τότε. Αλλά πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την αρχή της ίσης όλων των ομιλητών. Σας ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά για τις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ. Θέστε τις ερωτήσεις σας. Ή αν θέλετε τοποθετηθείτε σε κάποιο ζήτημα. Μόνο ενα θέλει το λόγο. Ο κύριος Στίβενσον. Μια ερώτηση για τον κύριο Μοντέρο. Για να δώσω και την ευκαιρία να, συνεχίσει αυτό το οποίο έλεγε. Η Πορτογαλία και ιδιαίτερα οι Αζόρες, την οποία την έχω επισκεφθεί επανειλημμένα, έχουν την, ε, ε, εμπειρία, τα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη των 200 μιλίων να πάει στα 100 μίλια χάρη ε, στην πολιτική ανοιχτή πρόσβαση στου κοινού πόρου. Ρωτώ, ε, αυτή η προσπάθεια πού οδήγησε. Οι βιοτέχνες αλληλείς βελτιώθηκαν, βελτιώθηκε η θέση τους, εξακολούθησαν να έχουν την ίδια επιτυχία. Και τι έγινε μετά από θέματα. Ε, από αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ. Κύριε Φράγκα. Ε, ε, ε, Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω ένα σχόλιο και μετά να κάνω μια ερώτηση και στους δύο μιλητές εκπροσώπους των κρατομελών. Να πω το εξή. Νομίζω ότι η ανάλυση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής δείχνει ότι έχει αποτύχει το μοντέλο διαχείριση. Και με εκπλήσει το γεγονό ότι εσεί επιμένετε για άλλη μια φορά προ την κατεύθυνση ενό μοντέλου που οι περισσότεροι, ο κλάδο κτλ. θεωρούν ότι, είναι, είναι, ότι έχει αποτύχει. Όσον αφορά την αρχή τη σχετική σταθερότητα. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα σα πω για τα προβλήματα, αλλά θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Η αρχή τη σχετική σταθερότητα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παραβιάζεται καθημερινά από τα κράτη-μέλη που προβαίνουν σε ανταλλαγέ ποσοστώσεων μεταξύ του κτλ. Άρα λοιπόν, να υποστηρίζετε μια αρχή που εσείς οι ίδιοι δεν τηρείτε, τι να σας πω, δεν, δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε. Και υπερασπίζεστε αυτή την αρχή η οποία δεν εφαρμόζεται μέσα από την καθημερινή πρακτική. Και δεύτερον, όσον αφορά τη Συμβουλευτική Επιτροπή, Καταλαβαίνω βεβαίω ότι εδώ εκφραζόμαστε διπλωματικά και με λεπτότητα όπως αρμόζει στις σχέσεις ε, ε, μεταξύ μα. Αλλά καταλαβαίνω ότι εδώ βρίσκεται το εξής παράπονο. Ότι δηλαδή δεν παίζουν ε, όπως θα έπρεπε το... δεν ασκούν όπως θα έπρεπε τη γνωμοδοτική του αρμοδιότητα τα ΡΑΞ. Και εγώ συμφωνώ όχι γιατί γνωρίζω ορισμένα τέτοια γνωμοδοτικά συμβούλια, αλλά και επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής παίζει γνωμοδοτικό ρόλο και όμως δεν μα δίνει και ιδιαίτερη προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε και το Συμβούλιο των Υπουργών. Άρα σα καταλαβαίνω πολύ καλά. Καταλαβαίνω την απογοήτευση που αισθάνεστε. Συν το γεγονό ότι πρόκειται για οργανισμού που ιδρύθηκαν πρόσφατα κτλ. Άρα, κάνω την εξή ερώτηση και είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριο Άντερσον. Το θέμα του ελέγχου. Το οποίο είναι σε μελιώδε. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση που γίνεται για του ελέγχου, τέλο πάντων δεν την κρίνω, αλλά είναι πολύ σημαντική και αφορά όλο τον τομέα. Α, επίσης θα ήταν πάρα πολύ καλό να εμπλακεί ο κλάδος και ο τομέας να είχε εμπλακεί κατά τη σύνταξη ε, τη πρώτη επιτροπή. Δηλαδή η επιτροπή να έχει ακούσει τι απόψει του τομέα. Γιατί αν δεν δεχθεί τι προτάσει περί ελέγχου ο τομέα, τότε δεν πρόκειται να εφαρμοστούν οι προτάσει αυτέ. Μιλάμε για ένα σύστημα που δεν είναι δυνατόν να το ελέγξουμε. Αν δεν το δέχεται και ο τομέα, τότε ε, εκ των προτέρων είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Ρωτώ. Παράδειγμα, τον εκπρόσωπο του, του, του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου έδωσαν την άποψή του για το θέμα του ελέγχου. Γνωμοδότησαν. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Mm. Ρωτώ λοιπόν, συμμετείχαν ε, στην συζήτηση, του ε, έλαβαν υπόψη την ε, θέση του. Αναφέρομαι και στον εκπρόσωπο του συγκεκριμένου ΡΑΚ, αλλά και στου υπόλοιπου. Κ. Καπούλα Σάντο. E eh, e, e- Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Κυρίως προς τον κύριο Ενρίκο Μοντέρο που έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αλίας. και γνωρίζει πολύ καλά την πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα μας. Λοιπόν, είπε ότι εδώ υπάρχουν μία σειρά από αρνητικές πτυχέ. Ε, μα αυτό είναι το θέμα. Μιλάμε και για τους πόρους και για την υπεραλίευση. Όλοι συμφωνούμε στη διάγνωση και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους η πολιτική αλίας με τόσο καλές αρχές και με τόσο καλά μέσα στην ουσία έδωσε πενιχρά αποτελέσματα, πολύ κάτω από τις προσδοκίες μας. Έθεσα μία ερώτηση προς τον Επιτροπό και να σου πω ότι δεν με ικανοποίησε η απάντησή του. Δηλαδή, η νέα προσέγγιση της Επιτροπής φαίνεται ότι στηρίζεται στην αρχή ε, διασφάλισης μίας σειράς προτεραιοτήτων. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και το θέμα των πόρων, το οποίο είναι θεμελιώδε σε όλη την προβληματική για την Ελία. Αλλά για να είναι διαρκής ε, η πόρη και επειδή υπάρχει υπεραλίευση, άμα δεν μειωθεί η υπεραλίευση, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για διατήρηση των αποθεμάτων. Αλλά αυτό σημαίνει απόλυτη θέση εργασία. Και μην ξεχνάτε, τα σημερινά οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια είναι ήδη πολύ δύσκολα. Και είναι δύσκολο για άτομα τα οποία δεν έχουν και πολλά προσόντα. Οπότε δεν έχουν και πολλέ δυνατότητε εξέβρεση άλλη απασχόληση. Γι' αυτό σα ρωτώ, δεν πιστεύετε ότι στο έγγραφο τη Επιτροπή εδώ υπάρχει ένα κενό πολύ σημαντικό που αφορά ε, τα μέτρα αποζημίωση έναντι των ανθρώπων αυτών που δεν έχουν άλλου πόρου και που θα χάσουν την εργασία του μέσα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε σε ερωτήσει αυτέ ε, που σα υπευλήθησαν. Muito obrigado. ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω με την ερώτηση με το θέμα των πλέον απομεμακρυσμένων περιφερειών. Ε, και ε, τέτοιο ερώτημα κατά πώς τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν άλλη δυνατότητα απασχόλησης και σε, σε σχέση και με τη μείωση της ζώνης αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης από τα 200 μίλια ε, οι Αζόρας και Μαδέρα πραγματικά είναι περιοχές οι οποίες ε, ζουν από την Αλία και πρέπει να προστατευτούν και οι οποίες καλύπτονται από το νέο αυτό όριο. Ε, ε, Τώρα η κυρία Φράγκα αναφέρθηκε στο θέμα σχετικής σταθερότητας. Χρειαζόμαστε πράγματι ένα μηχανισμό που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε, να κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει δηλαδή τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν ποσοστώσεις θέλουμε να βρούμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα μας εξασφαλίσει όταν θα διατηρηθεί η αληφτική δραστηριότητα εκεί όπου παραδοσιακά ε, είναι η κύρια σχολεία. Μοιραία λοιπόν πειραία λοιπόν η σταθερότητα πρέπει να εξασφαλιστεί και στο μέλλον. Επόμενη ερώτηση σχετικά με τη μείωση της δυναμικότητας και την, το πώς επηρεάζεται ε, ο ντόπιος πληθυσμός. Ρε εσύ Φωτεινή μπορείς να ακούς τα ισπανικά λίγο. Η εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια κάποια ιεραρχία. Θα πρέπει βεβαίως να εξασφαλίσουμε τα λευτικά αποθέματα, αλλά συγχρόνως να διατηρήσουμε και κάποιο κοινωνικό επίπεδο. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια κάποια, ένα κάποιο οικονομικό κέρδος αλλά η οικονομική και κοινωνική συνοχή είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια κάποια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε έτσι ώστε να υπάρχει απαραίτητη ισορροπία και πραγματική οικονομική και κοινωνική συνοχή. Όσον αφορά τα ζητήματα τα κοινωνικά, ε, η σημερινή ε, πολιτική έλαβε υπόψη την ε, πιθανή απώλεια θέσεων απασχόλησης, μιλά για ανάπτυξη ε, των παράκτιων περιοχών και δίδεται ε, βασικός ρόλος στις τοπικές αρχές που θα μπορέσουν να προτείνουν ε, ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης για να αντισταθμιστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας στην Ελία. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κανείς δεν τοποθετήθηκε στο θέμα αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να πω τα εξής πιστεύουμε ότι η διαχείριση των πόρων δεν είναι θέμα αποκλειστικά τεχνικό. Η αρχή της επικουρικότητας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση, ε, που, ε, τη βάση της διακυβέρνησης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις, οι θεμελιώδεις αποφάσεις, είτε όσον αφορά ε, το, το σεβασμό των βασικών ε, θέσεων ε, είτε τα βασικά ζητήματα πολιτικής πρέπει να λαμβάνονται από το Συμβούλιο με βάση την ισορροπία ανάμεσα στους διάφορους, ε, στα διάφορα επίπεδα ε, αποφάσεων. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, στην επόμενη ενότητα. Έχουμε τον κύριο Κάρλος Αλβερεγία ε, ο οποίος προέρχεται από το ΡΑΚ μεγάλης απόστασης, από την κυρία Τρουχιγιάνο, που προέρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Υπέθρου και και αλίας ε, τη Ισπανία και από τον κύριο Φραντσέσκο Αμπάτε, Γενικό Διευθυντή για την Αλία και την Ιχθυοκαλλιέργεια, από το Υπουργείο Γεωργίας Τροφίμων και Δασοκομεία τη Ιταλία. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Αλερεδεγία για 10 λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω είπατε και προηγουμένω, ε, δεν σα λέω ότι θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, θα είμαι. Λοιπόν, πριν από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελίας ε, του Κοινοβουλίου για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έρθω εδώ σήμερα και αντικαθιστώντας τον πρόεδρο του ε, Γνωμοτικού Συμβουλίου μας, ε, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει λόγω ε, ανηλυμένων υποχρεώσεων. Όπω ήδη αναφέρθηκε επανειλημμένα, ένα από τα βασικά επιτεύγματα τη μεταρρύθμιση τη κοινή ελευτική πολιτική του 2002 ήταν να συμμετέχει πολύ περισσότερο η κοινωνία των πολιτών αυτή η συμμετοχή και αυτή η μεγαλύτερη εμπλοκή υλοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας ε, των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, τα οποία έχουν βασική αποστολή να συμβουλεύουν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πτυχές της Ελίας που αφορούν τους δικούς τομείς αρμοδιότητας. Με την έννοια αυτή, ε, ε, το δικό μας ε, το ΡΑΚ ασχολείται με την αλία ε, εκτός των υδάτων δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Αυτό γίνεται με τρεις οδούς. Πρώτον, μέσω των συμφωνιών αλίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες, μέσω της συμμετοχής σε περιφερειακές οργανώσεις αλίας και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και τέλος μέσω ε, δράσεων που αφορούν την αγορά και το εξωτερικό εμπόριο στον τομέα της αλίας. Πρώτη οδός, ε, αλλιευτικές συμφωνίες. για πολλά χρόνια ε, ε συζητεί το θέμα και το 2003 το Συμβούλιο δημοσίευσε τις, τα συμπεράσματά του για τις ελευτικές αυτές συμφωνίες τονίζοντας το πόσο σημαντικές είναι οι συμφωνίες και εκεί αναφέρεται η βούληση διατήρηση των συμφωνιών αυτών ως θεμελιώδες στοιχείο της ε, κοινής ελευτικής Ανάμεσα στα ε, τονίζουμε το, την οικονομική αντιστάθμιση που ε, μαζί με άλλα θέματα όπως ε, φορολογία, τέλη, λιμενικά κτλ. Όλα αυτά όλα αυτά είναι πάρα πολύ, ε, ένα μεγάλο βάρος του ΑΕΠ των τρίτων χωρών. Μέσω όμω τη συνεργασία ε, στην ανάπτυξη ε, μπορεί να βρεθεί λύση και σε όλα αυτά τα ζητήματα. Πέραν τούτων όμω, ε, τα, τα κοινοτικά πλοία τα οποία αλλιεύουν στι τρίτε χώρε έχουν πλήρωμα τοπικών πληθυσμών. Άρα σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και η μετανάστευση των ανθρώπων αυτών εφόσον βρίσκουν εργασία επιτόπου. Πρέπει να δούμε όμως τώρα ότι ό,τι αφήνουν ε, τα κοινοτικά πλοία καλύπτεται από παράνομη αλεία. Και με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η ανάπτυξη και των τοπικών ε, στόλων. Εμείς λοιπόν εκ μέρους του Συμβουλίου μας ζητούμε η νέα ε, ε, πολιτική να ε, προωθήσει ε, ακόμα περισσότερο την αλληλεία των πλοίων στα, στα τα αυτά δικαιοδοσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην διατηρώντας αυτά που υπάρχουν και στην εξέβρεση νέων λύσεων. Όσον αφορά τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας, εδώ πρέπει να πούμε ότι το μέλλον των, ε, των οικονομικών πόρων περνά μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση. Με αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ε, ιδιαίτερη δραστηριότητα σε αυτές τις οργανώσεις και ε, ζητάμε να εξακολουθήσει να παίζει καθοδηγητικό ρόλο σε αυτές τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας. Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι, ότι τα μέτρα διαχείριση είναι ευθύνη τόσο των χωρών παραγωγή αλλά και των χωρών στι οποίε γίνεται η εμπορία. Εδώ η κοινοτική δράση ήταν ιδιαίτερα έντονη και όλα αυτά είναι ουσιαστικά ε, για την ε, καταπολέμηση ε, της παράνομης αντίληψης και ανεξέλεκτης ελίας. Πρέπει να προωθήσουμε την, τη συνεργασία των περιφερειακών οργανώσεων αλίας με τις χώρες με τις οποίες υπάρχουν αλληλευτικές συμφωνίες για να προωθήσουμε το διάλογο σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τη δραστηριότητα των δικών μας τόλων σε αυτά τα ύδατα, εδώ σα επιστώ την προσοχή σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα μέλη της Επιτροπής μας, που είναι το θέμα ε, της πειρατεία. Όπως όλοι γνωρίζετε, η κατάστασή του τελευταίους μήνες είναι αβάσταχτη. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους του, όλα τα όργανα, όλων των κρατών μελών, ε, όλους τους θεσμούς για τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει μέχρι στιγμής. Και σας παρακαλούμε να ε, ε, ε, βοηθήσετε τα πλοία και να τους βοηθήσετε έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια. Τρίτη οδός που αφορά τις δράσεις που αφορούν την, ε, ε, την αγορά και το εξωτερικό εμπόριο. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μία από τους, βασικές, από τους βασικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο των αλλιευτικών προϊόντων. Άρα πρέπει η πολιτική αγοράς να συμβαδίζει με την αλλιευτική πολιτική. Να εγκριθούν μέτρα τα οποία να βοηθούν τους νόμους και να τιμωρούν τους παράνομους. Και με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε και το θέμα της αποφυγής της παράνομης αλίας. Τώρα, ε, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν το πόσο σημαντική είναι η διεθνή διάσταση, η εξωτερική διάσταση αλληλεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 720 κοινοτικά πλοία τα οποία αλλιεύουν σε διεθνή ύδατα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από μία έκθεση ε, την οποία την αφέσαμε σε εξωτερικό γραφείο συμβούλων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη αυτή και μπορείτε να τη δείτε και στην ιστοσελίδα μα. 720 πλοία λιγότερο για το 1% του κοινοτικού στόλου, αλλά το 24% τη ολική χωρητικότητας και το 9% των κιλοβάτ. Ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο άρθρο 39 της συνθήκης, εκεί όπου ορίζονται οι στόχοι της κοινή ε, πολιτικής του τομέα της αναφέρεται και ε, η αυτάρκη εφοδιασμού. Και εδώ μιλάμε για 1,2 εκατομμύρια τόνους, το 21% ε, του συνόλου της αγοράς της κοινοτικής, πάντα για τα προϊόντα αλίας. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν αντικατοπτρίζουν ε, ε, το πόσο σημαντικό είναι ο στόλο αυτό που ελιεύει στα διεθνή ύδατα. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στη νέα μεταρρύθμιση τη κοινή πολιτική στον τομέα τη ελεία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μείνατε ε, μέσα στο χρόνο σας, ε, τηρήσατε το λόγο σας, είπατε θα είμαι σύντομος και ήσασταν σύντομος χαρτήρια Να δώσω το λόγο λοιπόν στην επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, ε, να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δώσατε να έρθουμε εδώ ε, στην ακρόαση αυτή και να συζητήσουμε ένα θέμα τόσο σημαντικό. Φάνηκε το πόσο σημαντικό είναι από τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ομιλητών και το ενδιαφέρον το οποίο παρουσιάζει. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο ο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα και πολύτιμο, θα ε, αναφερθώ κατευθείαν σε ορισμένες βελτιώσεις που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτα απ' όλα λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ε, κατάσταση στην κοινή ελευθερική πολιτική και να δούμε την μελλοντική κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για, ε, ορισμένες, για την πρόοδο που υπήρξε και που την τόνισαν και ορισμένοι από τους προλαλήσαντες, όπως για παράδειγμα όσον αφορά τα σχέδια μακροπρόθεσμης διαχείρισης, την, τώρα τότε στηριζόμαστε στη μέγιστη απόδοση, ε, διαρκή απόδειξη ε, στην, ε, στην προσέγγιση την οικοσυστημική, στην βελτίωση της κυβέρνηση, στην βελτίωση της επιστημονικής ενημέρωσης κτλ. Όμως, σε κάθε, ένα από τις, σε κάθε μία από τις στοιχείες αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία και πτυχές στις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στην ιδανική κατάσταση. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείριση, εξακολουθεί να λείπει η βιολογική μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Τα, ε, τα βραχυπρόθεσμα σενάρια πολλέ φορέ εμπεριέχουν δραστικά κοινωνικο-οικονομικά μέτρα, τα οποία είναι δύσκολο να αναλυφθούν. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό που λείπει είναι κάποιοι προσανατολισμοί διαχείριση, περισσότερο μακροπρόθεσμοι, με ενδιάμεση αναθεώρηση, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει ο τομέα ε, να μπορέσει να τα αφομοιώσει αυτά τα σχέδια και να τα εφαρμόσει αυτά τα σχέδια ε, με καλύτερο τρόπο. Διότι και από βιολογική άποψη θα είναι καλύτερα, αλλά και ε, θα παρουσιάζουν λιγότερο άχθο από οικονομική άποψη. Μιλάμε επίση για τη μέγιστη διαρκή απόδοση. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τον ορισμό. Δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε στην τιμή της ε, θνησιμότητας ε, αυτό που ονομάζουμε FM-SY όταν πρόκειται ε, για ε, αλληλεία διαφόρων ειδών. Δηλαδή, ε, είναι ε, η θνησιμότητα ε, του πλέον αλλιευμένου είδους αυτού που, που οδηγεί σε λιγότερη απόδοση. Καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για αλλία ενός και μόνο είδους δεν έχουμε πρόβλημα. Όταν όμως μιλάμε για αλλίες πολλών ειδών δεν έχουμε καταφέρει για ποια θνησιμότητα ανά αλλία μιλάμε. Πράγμα το οποίο αποτελεί επιθυμητό στόχο. Μιλάμε για απορρίψει. Ωραία, όλοι συμφωνούμε. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να καταργηθεί αυτό το φαινόμενο. Αλλά σα ευχαριστώ την προσοχή στο γεγονό ότι μερικέ φορέ οι απορρίψει Μάλιστα, μιλάμε πάντα για επιλεκτικότητα, αλλά δεν έχει πάντα σχέση το πρόβλημα αυτό με την επιλεκτικότητα. Πολλέ φορέ οι απορρίψει γίνονται λόγω έλλειψη ε, ποσόστοση. Ή επειδή δεν υπάρχουν ή επειδή έχουν εξαντληθεί οι ποσοστώσεις. Τώρα, όσον αφορά την ε, οικοσυστημική προσέγγιση, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Επίτροπο, εδώ έχουμε διάφορε κατευθύνσει που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλε οι οικονομικέ δραστηριότητε που αναπτύσσονται στον κόσμο τη θάλασσα, στα διεθνή πλαίσια επίση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μιλάμε για τη διακυβέρνηση, θέμα στο οποίο επίση αναφέρθηκαν και άλλοι ομιλητέ που πήραν το λόγο προηγουμένω. Πρώτα απ' όλα όμω θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε να ξεκαθαρίσουμε και να διατηρήσουμε τη σημερινή ισορροπία αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Επίση, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, όλοι αναφερόμαστε στη, δημιουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων και στη λειτουργία του. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα ΡΑΞ, και εγώ πιστεύω θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά τη λειτουργία τους οι δομέ του διακυβέρνηση μερικέ φορέ είναι ιδιαίτερα άκαμπτε, να το λάβουμε υπόψη, και παρουσιάζουν την εξή δυσκολία. Να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε τον τομέα της αλίας, της παραγωγής, της βιομηχανίας και μερικές φορές ε, όλοι αυτοί οι κλάδοι δεν, δεν έχουν την ίδια προσέγγιση και δεν ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία. Λαμβάνοντα υπόψη την ίδια δυναμική επεξεργασία των κανόνων, αναφέρθηκε πολλέ φορέ ότι μερικέ φορέ γνωμοδοτεί το για ένα συμβούλιο, για ένα θέμα, συγγνώμη, το οποίο συζητά το Συμβούλιο. Μα τι αρμοδιότητα γνωμοδότηση έχει το ΡΑΚ, ήδη, όταν ήδη το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε επίπεδο Συμβουλίου. Ε, μα και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το αναλύσουμε. Άλλε πτυχέ. Ε, Λεπτομέρειε, αλλά πολύ σημαντικέ. Ε, ε, κοιτάξτε, όσον αφορά ε, τη, ε, τη γλώσσα εργασία. Υπάρχουν χώρε, τι οποίε πολλέ φορέ τα έγγραφα φτάνουν με δύο ή τρει εβδομάδε καθυστέρηση έναντι του πρωτότυπου. Ακριβώ γιατί απαιτείται μετάφραση. Μα αυτέ οι δύο ή τρει εβδομάδε ε, τις εκμεταλλεύονται ορισμένοι για να προχωρήσουν ενώ άλλοι δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν. Είναι λεπτομέρειες όλα αυτά, είναι και απλά πράγματα ε, και τα οποία ε, δείχνουν ότι δεν, δεν δουλεύουμε όλοι κάτω από ισότιμες ε, συνθήκες. Επίσης, επιστημονικά στοιχεία και ποιότητά τους αναφέρθηκα ε, επίσης ε, στο γεγονός ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει περισσότερο ο αλληλευτικός τομέας ε, το τι γίνεται. Αλλά εκεί όπου αντιμετωπίζουμε τις περισσότερες δυσκολίες κατά την άποψή μου είναι το θέμα των τάκ και ποσοστώσεων. Κατά την άποψή μου το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα άκαμπτο, στηρίζεται σε μία αρχή που δεν είναι επικαιροποιημένη που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα του αλληλευτικού τομέα και με των ανθρώπων που ζουν από την αλλία που δεν ικανοποιεί ούτε τον αλληλευτικό κλάδο, ούτε τις διοικήσεις, ούτε τους επιστήμονες και που αποτελεί αντικείμενο σταδιακών μειώσεων για επιστημονικού λόγου σε κοινοτικό επίπεδο, σε διεθνέ επίπεδο, είτε πρόκειται για τη, μέγιστη, για τη μέγιστη απόδοση, είτε για την οικοσυστημική προσέγγιση και μερικέ φορέ επειδή πρόκειται για αυτό που λέμε paper fish. Μερικέ φορέ, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία βεβαίω και δεν μπορούν να βελτιωθούν, ο ΑΛΙΕΦ αυτό το οποίο βλέπει είναι τη μείωση των αλληλευτικών του ε, ε, δυνατοτήτων και αισθάνεται απειλή. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα με ποσοστό, όσον αφορά ορισμένα αποθέματα και ορισμένε χώρε. Η ανταλλαγή ποσοστώσεων, θέμα στο οποίο επίση ε, αναφερθήκαμε εδώ, τα swaps, δεν λύνουν το πρόβλημα τη έλλειψη των ποσοστώσεων. Το ρυθμίζουν κάπω αλλά δεν το επιλύουν. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώνεται όταν τα τάκ κατα, ορίζονται σε επίπεδο αλλιεύματο. Δηλαδή όταν θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αυξηθούν σε επίπεδο αλλιεύματο, τότε αυτό ορίζεται ω οροφή. Αλλά υπάρχει και το εξή πρόβλημα. Ε, έχουμε ε, πλεόνασμα ποσοστώσεων που δεν τι εκμεταλλεύεται κανείς. Και κλείνουν ε, ε, κλείνουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ελεία συγκεκριμένων ειδών. Άρα σε τελευταία ανάλυση εξακολουθούμε να έχουμε τη βιολογική ζημιά και από την άλλη ε, δεν υπάρχει αλία. Πολύ σύντομα τα είπα όλα αυτά ε, για να σας δείξω και, και μάλιστα ε, πέρσι προετοίμασα εγώ μία μελέτη σε σχέση με τα αποθέματα του μπακαλιάρου του, του, του, του, Βορρά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τραντικού για την, σημαντικό είδος για την Ισπανία. Κάνα μία μελέτη στο διάστημα από το 2000 2006 και είδαμε τα αποθέματα που μένουν χωρίς αλία στη θάλασσα. Το 2001 1,6 ε, ε πάντων 26,9 το 2006 και ε, φτάνουμε στην κατάσταση των τεσσάρων αποθεμάτων ε, που συνιστούν τα αποθέματα του συγκεκριμένου είδους. Το κίτρινο τμήμα είναι αυτό το οποίο αλλιεύεται και το πράσινο είναι αυτό το οποίο δεν αλλιεύεται και μένει στη θάλασσα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι είναι, πάρα είναι κάπως δύσκολο να καταλάβουν οι αλλοίες τι γίνεται. Από τη μια κλείνουν λόγω έλλειψη ποσοστώσεων ε, οι, αλλη, τα, ε, οι επιχειρήσεις ορισμένε χώρε και από την άλλη παραμένουν από θέματα που δεν αλλιεύονται στη θάλασσα. Και επίση, να σα πω δύο λόγια. Όσον αφορά πάλι το κλείσιμο των επιχειρήσεων και τι επιπτώσει. Πολύ σύντομα θα σα πω το εξή. Θέλω να σα δείξω ότι, για παράδειγμα, το 2008 το 23,4 των αποθεμάτων ε, έκλεισε πριν φτάσουμε στο τέλο του χρόνου. Δηλαδή ε, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν φτάνει καν στο τέλος του χρόνου. Αν αυτό το λάβουμε υπόψη. Όχι μόνο. Και το συγκρίνουμε και με τον αριθμό των χωρών ε, όπου κλείνουν τα αποθέματα αυτά, σας λέω ότι βρισκόμαστε στο 37%. Θα πάμε στο 37%. Και αν δούμε τι γίνεται με τα βυθόβια ήδη, εκεί καταλαβαίνετε ότι το να κλείνουν επιχειρήσεις πριν τελειώνει το χρόνο, φτάνουμε στο 50%. Αυτά για το 2008. Καταλαβαίνετε πάντως ότι είναι αριθμοί ε, που μιλούν από μόνοι τους. Λοιπόν, οι ποσοστώσεις δεν είναι πανάκια. Γιατί δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Μια λύση λοιπόν θα μπορούσε να είναι η αλευτική ικανότητα. Και η αρχή που θα μας καθοδηγήσει για την επόμενη μεταρρύθμιση να είναι η αλληλευτική ικανότητα τα 15 δευτερόλεπτα που απομένουν θα ήθελα να τα αφιερώσω στο εξή. Να ε, σας ε, ε, πω δύο λόγια για την εξωτερική πολιτική όπου πιστεύω ότι τόσο όσον αφορά το θέμα ε, της ε, εργασίας περιφερειακές αλλά τόσο σε επίπεδο συμφωνιών, θα πρέπει και στο μέλλον να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Διότι ε, είναι πολύ σημαντική η εξωτερική διάσταση της αλίας. είναι και εκτιμένο, το οποίο δεν πρέπει να το χάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία μου και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φραντσέσκο Σαβερίο Αμπάτε, Γενικό Διευθυντή για τα Ελευτικά Ζητήματα από το Ιταλικό Υπουργείο Υπέθρου Τροφίμων και Δασοκομεία. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μερικέ φορέ το να παίρνει κανεί το λόγο τελευταίο αντιμετωπίζει δυσκολίε γιατί από τη μια ίσω επαναλάβει ορισμένα πράγματα τα οποία ελέγχθησαν και προηγήθηκαν ορισμένε παρατηρήσει. Βέβαια, πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή Αλία ε, για την σημερινή ακρόαση, για την κατάσταση ε, τη κοινή πολιτική δομέα τη Αλία και τι προοπτικέ. Σε ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή, για την πρόσκληση που μα απευθύνεται. Όπω είναι γνωστό, η, η βασική νομοθεσία, ο κανονισμός 2371-2002, δεν καθορίζει καμία προθεσμία για την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και δεν προβλέπεται ούτε καν, όπως όλοι γνωρίζουμε, ε, ενδιάμεση επανεξέταση. Πράγματι, η μοναδική υποχρέωση που αναλαμβάνει το Συμβούλιο είναι η επανεξέταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 των διατάξεων που περιέχονται στο άρθρο 17 και που αφορούν τις λεπτομέρειες πρόσβασης στα ύδατα τα οποία βρίσκονται μέσα στα 12 μίλια ε, από τις ακτές των κρατών μελών. Όμως ε, η Ιταλική κυβέρνηση ε, υποστηρίζει τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει για την προετοιμασία μιας νέας μεταρρύθμισης κοινή πολιτικής στο τομέα της Αλίας μετά από αυτή που αποφάσισε το Συμβούλιο 2002. Επιτρέψτε μου όμως ε, και εγώ να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά αυτά τα οποία πρέπει να περιέχει η κοινή αλληλευτική πολιτική. Κατά την άποψή μας, τα αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν είναι στο σύνολό του θετικά. Υπάρχουν σαφείς και ενισχυτικές ελλείψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκε η Επιτροπή, το 30% των αποθεμάτων για τα οποία υπάρχουν επιστημονικές πληροφορίες έχουν υπερβεί τα βιολογικά όρια ασφάλειας. Η οικονομική κατάσταση των ελευτικών επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιητική και η πρόσφατη κρίση ε, των τιμών ε, των καυσίμων τα περασμένα χρόνια, που όπως όλοι γνωρίζουμε και μέσα από τις ανησυχητικές εκδηλώσεις που έγιναν, ε, δημιούργησαν ακόμα περισσότερες δυσκολίες. Όμως η Ιταλική κυβέρνηση δεν συμφωνεί με ορισμένες αξιολογήσεις και ορισμένες αναφορές του εγγράφου που ε, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου του 2008 εν ώψη του άτυπου συμβουλίου που διοργάνωσε η Γαλλική Προεδρία. Σύμφωνα με την ανάλυση τη Επιτροπή, η κρίσιμη κατάσταση των αποθεμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τι επιλογέ που έγιναν από το Συμβούλιο, το οποίο στο πλαίσιο των ετήσιων αποφάσεων για τα μέγιστα όρια ε, προ, ε, προώθησε ε, βραχυπρόθεσμες λύσεις αντί να ε, προωθήσει ε, μακροπρόθεσμες λύσεις και βιώσιμες. Υπογραμμίζω αυτή εξ αρχή ότι οι ποσοστώσει ελευμάτων δεν αφορούν στον ίδιο βαθμό όλα τα κοινοτικά ύδατα. Για το λόγο αυτό, οι, οι, οι κριτικέ μα δεν μπορεί να είναι γενικευμένε. Όσον αφορά την αλληλεία στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, υπάρχει μία και μόνο ποσόστοση που αφορά τον ερυθρό ε, τόνο ε, και η οποία μειώνεται ακόμα περισσότερο λόγω των, των θέσεων ε, τη Διεθνού Επιτροπή για την Προστασία του Τόνου του Ατλαντικού. Όπω ήδη αναφέρθηκε ε, και μάλιστα πρόσφατα στι 29 Σεπτεμβρίου 2008 από την Ιταλική ε, Αντιπροσωπεία στο Άτυπο Συμβούλιο ευρύτερη προσφυγή εκ μέρου τη Επιτροπή ε, στα μέσα που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία θα είχε οδηγήσει σε καλύτερη προστασία των πόρων. Η αναφορά είναι, σαφ... Ε, είναι σαφές ότι η αναφορά ε, στα επίγοντα μέτρα όπως προβλέπονται από το άρθρο 7 του κανονισμού 2371 όταν παρουσιάζεται σοβαρός κίνδυνος για την διατήρηση των, των πόρων. Με βάση όλα αυτά, η Ιταλική κυβέρνηση θέλει να υπογραμμίσει δύο σημεία τα οποία, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ σημαντικά, λαμβάνοντα υπόψη την προοπτική μεταρρύθμιση τη κοινή ε, πολιτική στον τομέα τη Ελία. Πρώτα απ' όλα, ε, πρέπει να απλοποιηθεί ε, η υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη τόσο για τι εθνικέ κυβερνήσει, όσο και για του εκπροσώπου του κλάδου. Δεύτερον, αποκέντρωση των αποφάσεων. Τα τελευταία χρόνια έγιναν, αυτό είναι αλήθεια, σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την προετοιμασία των αποφάσεων του Συμβουλίου στο τέλος του έτους για τα μέγιστα επίπεδα ε, αλίας και για τα συναφή μέτρα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά ακόμα. Ένα και μόνο παράδειγμα θα σας ε, θέσω για να καταλάβουμε το πόσο ε, περίπλοκη είναι η νομοθεσία. Για παράδειγμα, η, νομοθεσία, ε, ε, η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει σχέδια αναδιάρθρωση, σχέδια ανάκτησης μακροπρόθεσμα, σχέδια διαχείριση σε κοινοτικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα σχέδια, τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ του, όλα οδεύουν προ την ίδια κατεύθυνση. Διατήρηση και προστασία των αποθεμάτων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Με την προσαρμογή της ελευτική προσπάθεια, προσαρμογή λοιπόν τη ελευτική προσπάθειας στην κατάσταση των αποθεμάτων. Δεύτερο σημείο αποκέντρωση των αποφάσεων. Για το θέμα αυτό θα πρέπει να εμβαθύνουμε την εξέταση ενός συστήματος για την προστασία των πόρων, το οποίο να είναι πιο ευέλικτο και να προσαρμόζεται καλύτερα στις διάφορες ε, τοπικές πραγματικότητες. Βεβαίως να είναι συνεπές και σύμφωνο με τους πολιετή στόχους που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και προωθώντας όλο και περισσότερο το ρόλο των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων. Θα θέλαμε τώρα να τονίσουμε ε, να, να, να επιστήσουμε την προσοχή σας σε δύο άλλες πτυχές. Πρώτα απ' όλα ε, όσον αφορά ε, την, την απόσυρση των σκαφών, τη διάλυση των σκαφών. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί το βασικό στόχο και της μελλοντικής πολιτικής στον τομέα αυτό. Τα τελευταία 15 χρόνια η ικανότητα του κοινοτικού στόλου μειώνεται κάθε χρόνο κατά 1,5%. Ε, και ε, ε, κατά 1,5% όσον αφορά τη χωρητικότητα και κατά 2% όσον αφορά την ισχύ τη μηχανή. Παρά την ένταξη νέων κρατών μελών το 2004-2007, σήμερα ο ε, στόλος είναι, είναι μικρότερος κατά 18.000 μονάδες έναντι του επίπεδου του 95. Καταλαβαίνετε λοιπόν το κοινωνικό κόστος αλλά και το οικονομικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξέταση σε βάθος. Για μας ε, θα ήταν χρήσιμο ε, στο μέλλον να αναλάβει σημαντικό ρόλο, ε, να είναι πολύ πιο σημαντικός ο έλεγχος αλληλευτικής προσπάθεια που θα γίνεται μέσα από προσωρινή πάυση των δραστηριοτήτων και προγραμματισμένη. Το άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ στα λίγα λεφτά που μου απομένουν αφορά την ε, κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα ε, της κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής. Στο έγγραφο το οποίο σας ανέφερα πριν από λίγο και που έχει ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή ανέφερε ότι η οικολογική βιωσιμότητα είναι βασική και έχει προτεραιότητα έναντι τη κοινωνική και τη οικονομική. Ήδη στο άτυπο συμβούλιο η Ιταλική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τη θέση αυτή διότι πίσω από την κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα βρίσκεται η απασχόληση και τα έσοδα πολλών οικογενειών και επιχειρήσεων. Άρα το θέμα αυτό θα πρέπει να, να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ε, τώρα, φτάνω στα συμπεράσματα και θα ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι κάτι το, ε, ε, που δίνει ιδιαίτερη σημασία ο κλάδος μας αλίας. Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα έναν των τρίτων χωρών. Σας υπενθυμίζω, το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε αλλιευτικά προϊόντα ε, ύψους 16 δις ευρώ. Στι αρχέ τη δεκαετία του 70, η εσωτερική κατανάλωση καλυπτόταν κατά 75% από προϊόντα τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο αλλία. στα κοινοτικά ύδατα. Το ποσοστό αυτό τώρα έχει μειωθεί στο 40%. Οι επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τι τρίτε χώρε. Και υπό την οπτική αυτή γωνία έχουμε συγκεκριμένε ε, ευθύνε. Όμω θα πρέπει να καταλάβουμε τι ε, συνέπειε που έχουν οι αποφάσει μα ε, ω προ την προστασία των αποθεμάτων. Για παράδειγμα, να, πάρουμε, να δούμε τι γίνεται με την αλία στη Μεσόγειο ε, με βάση τα τελευταία στοιχεία που εξεργάστηκε η Επιτροπή, από το 1992 στο 2005 τα αλλιεύματα από τον κοινοτικό στόλο μειώθηκαν κατά 22%. Ενώ τα συνολικά αλλιεύματα μειώθηκαν μόλις κατά 1%. Στην ουσία, ε, το, το πεδίο ε, που άφησε ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύφθηκε από άλλες χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πίεση στα αποθέματα παρέμεινε ίδια ουσιαστικά. Τέλο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε ένα θέμα το οποίο αφορά την εμπορία των αναλυτικών προϊόντων. Ο ρόλο των οργανώσεων των παραγωγών περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, για να μην πούμε ότι έχει εκμηδενιστεί, από την διαχείριση τη προσφορά και κατά συνέπεια ε, τη ε, διαδικασία διαμόρφωση των τιμών είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι αλήθεια. Στα πλέ, Και θα το εξετάσει στα πλαίσια τη επόμενη αναθεώρηση τη κοινή οργάνωση αγορά. Όμω ο στόχο τη καλύτερη εμπορία και αξιοποίηση των προϊόντων θα πρέπει να έχει προτεραιότητα και, στις, ε, ε, ε, και στον προβληματισμό που έχει να κάνει με την αναθεώρηση τη κοινή αλληλευτική πολιτική πιο ικανοποιητική ε, ε, και σταθερή αποδοτικότητα ε, θα οδηγήσει στο να αλληλείς στο να περιορίσουν τις ημέρες αλίας και τις ημέρες των ημερών στη θάλασσα. Τελειώνω λέγοντάς σας ότι η επόμενη κοινοτική πολιτική στον τομέα της αλίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία αλλά να υποστηρίζεται και από τους κατάλληλους πόρους στη, στην περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Μπάτ, Δεν μου έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Φράντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία σειρά από ερωτήσει στους, ε, δύο ε, προσώπους των ε, ΡΑΚ σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρει το έγγραφο της Επιτροπής για την Εξωτερική Πολιτική και για τις ε, αλληλευτικές συμφωνίες. Όταν αναφέρεται η φυστάμενη κατάσταση, και θέλω να πείτε αν συμφωνείτε, γιατί εγώ δεν συμφωνώ, αναφέρεται ότι οι, οι ευρωπαϊκοί στόλοι εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δημόσιες ενισχύσεις για να λιεύουν στα, στα διεθνή Μα εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Μόνο από τη, από τις, ε, από τη δημόσια ε, βοήθεια και ενίσχυση εξαρτώνται. Και κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει Ε, αναφέρεται ε, σε μια συγκεκριμένη αντίληψη που έχει για την ικανότητα αλλιευσής στα διεθνή ύδατα. Ρωτώ, είναι γενικευμένη η άποψη αυτή ή αφορά μόνο την άποψη ενός συγκεκριμένου τμήματος της κοινωνία. Και επίση, όσον αφορά την προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι συμφωνίε που αφορά αποκλειστικά, τουλάχιστον έτσι γράφει το έγγραφο, έτσι γράφεται στο έγγραφο ε, στο θέμα ε, της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη, όχι στο θέμα των αλληλευτικών σχέσεων. Και κάτι άλλο. Στα μέλη σας, στο δικό σας το ΡΑΚ, τι εντύπωση επικρατεί ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στο θέμα καταπολέμησης της αδήλωτης, ανεξέλεγκτης και παράνομης αλίας. Και να πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά το θέμα της υπεραλίευσης να κάνετε ψυχόλιο. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Εντάξει, ακούσαμε όλα αυτά που ακούσαμε για το μοντέλο διαχείρισης, το οποίο... Α, κυρία Φράγκα, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Ε, ε, όχι, εντάξει, λέει κυρία Φράγκα, τελειώνω. Γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως βλέπετε, λέει η πρόεδρος, δεν έχουμε χρόνο. Ε, μα και εγώ θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, λέει η πρόεδρος. Ρωτώ, λέει η κυρία Φράγκα, ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο επίτροπο και με τον νέο κανονισμό ε, για τη διαχείριση κρίσης, ε, το οποίο συνεκρίθη, και με τι πιθανέ ενισχύσει για 700 εκατομμύρια ευρώ για φέτο και για τα επόμενα χρόνια. υπάρχει εντύπωση ότι αυτός ο μηχανισμός δεν αντιμετωπίζεται καθόλου. Μα εγώ ξέρω ότι σε ορισμένα κράτη, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, ζητήθηκαν πολλά χρήματα για τη διάλυση και δεν έγινε τίποτα. Άρα λοιπόν θέλω να μάθω είναι γενικευμένη αυτή η στάση ή τι γίνεται, γιατί εδώ μας, ε, ε, ε μας ζητάτε βοήθεια, όλοι εργαζόμαστε και μετά λέτε δεν κάνουμε τίποτα. Ε, θέλω λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σας. Κοιτάξτε. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής που θέλει να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις. Αλλά να, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Εγώ χθε συμμετείχα σε μια συνεδρίαση από της Υποεπιτροπής Άμυνας για να μιλήσουμε για το πρόβλημα της Σομαλίας και την πειρατεία. Και τι είδα. Τρει από του εκπροσώπου τη Επιτροπή ε, που συμμετείχαν, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συμμετείχαν στην συνεδρίαση αυτή, από τη Γενική Διεύθυνση Συνεργασία για την Ανάπτυξη, μίλησαν για την υποτιθέμενη παράνομη αλία στα ύδατα της Σομαλίας που ήδη με εξέπληξε και συνέδεσαν το φαινόμενο αυτό με το φαινόμενο της ε, πειρατείας επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω έτσι αυτές, ε, αυτή τη δημιουργία εντυπώσεων ότι η Σομαλία δηλαδή υπάρχει πειρατεία λόγω της παράνομης ε, αλίας και κατά κάποιο τρόπο η πειρατεία είναι απάντηση σε αυτές τις δραστηριότητες παράνομης αλίας και επειδή δεν καταδεικνύεται καμία χώρα. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η υπόνοια αφορά όλες τις ε, χώρες και τις χώρες, μέλη. Ρωτώ τον κύριο Δεμπέν. Η Γενική Διεύθυνση Αλίας έχει συνειδητοποιήσει ότι ότι, αυτοί, ε, ότι αυτοί, αυτές οι υπόνοιες εξαπλώνονται. Εσείς με βάση τις, τις συνεδριάσεις που κάνετε για, την, για το φαινόμενο της πειρατείας στη Σομαλία έχετε να μας πείτε κάτι τέτοιο και μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα έγγραφο το οποίο να εξηγεί σε τι συνίσταται η δραστηριότητα των κοινοτικών πλοίων που ελιεύουν στα διεθνή ύδατα και συγκεκριμένα στις ακτές της Σομαλίας. Ίσως αυτό ήταν πιο πρακτικό. Ε, σας δίνω το λόγο. Πολύ σύντομα να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ δεν ήμουν σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά το μόνο που θα σα πω είναι ότι η επίσημη θέση τη Επιτροπή και στη συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση για τι Θάλασσε είναι ότι δεν συσχετίζεται καθόλου η δραστηριότητα του κοινοτικού στόλου ε, στα ύδατα τη Σομαλία με την ανάπτυξη τη πειρατεία. Από την άλλη μεριά να σα πω ότι η πειρατεία δεν αφορά ιδιαίτερα τον κοινοτικό στόλο, ε, αφορά ε, τα πετρεολεοφόρα, την ανθρωπιστική βοήθεια, όλου του στόλου. και όλο τα είδη πλοίων. Δεν νομίζω ότι είναι σωστέ αυτέ οι αναλύσει, είναι υπερβολικέ. Θα ρωτήσω όμω από του συναδέλφου να μου πούν πού στηρίζονται. Όσον αφορά τη θέση τη Επιτροπή, είναι σαφέστατη. πάντα υποστηρίζαμε ε, ε τι προσπάθειε προ την κατεύθυνση αυτή. Ε, χρηματοδοτήσαμε τι μελέτε ε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση μα είναι σαφή. Ε, άμεση στήριξη σε αυτό το σύστημα πρόληψη πειρατεία. Όσον αφορά τη συζήτηση διμερινή, κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, πάρα πολύ σύντομα, μα δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα σχόλια τα οποία έγιναν μέσα σε τόσα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μα. Απλά και ε, να, να, να, να μεταφέρω δύο μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, ακούσαμε τον κύριο Σου ότι συμμετείχε στι συζητήσει του 1992, του 98 και του 2002. Μα νομίζω ότι και άλλα μέλη τη Επιτροπή σα ε, συμμετείχαν σε αυτέ τι συζητήσει. Εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να το πράξω, αλλά όταν ο Επίτροπο μα ανέθεσε ε, να μελετήσουμε τη μεταρρύθμιση, μελετήσαμε όλα τα έγγραφα από το 1992, το 98, το 2002. Είδαμε όλες τις διαδικασίε ε, μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτική ε, πολιτική. Μέσα από όλα αυτά τα έγγραφα και εκεί παντού οι αναλύσεις είναι οι ίδιες. Τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι τα ίδια. Ε, το διακύβευμα, οι δεσμεύσει, οι λύσει είναι ίδιε. Οι κριτικέ, οι ίδιε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που θα πρέπει να θέσουμε σε αυτή την έναρξη του προβληματισμού είναι η εξή. Γιατί αποτύχαμε, Γιατί στι τρει τελευταίε μεταρρυθμίσει, ενώ λέμε τα ίδια, δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Και ίσως η απάντηση είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές έγιναν με βάση μιας λογικής του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Ε, του συμβιβασμού ανάμεσα σε όλους. Και αυτό δεν μας οδήγησε πουθενά. Αυτό πρέπει να δούμε. Παρουσια... Δώσαμε σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, ένα πρώτο γύρο διάγνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις, ε, βασικές βασικέ τοποθετήσει μα που δικαιολογούν το να γίνει νωρί, όσο αυτό νωρίτερα η μεταρρύθμιση. Υπάρχει γενικευμένη συνένεση. Κανένα Κανένα κράτος-μέλος δεν διαφώνησε όσον αφορά τη διάγνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικά. Τώρα, σαν πρώτη λεπτομέρειε, εντάξει, αλλά η διάγνωση είναι η ίδια, η διάγνωση είναι κοινή. Δυστυχώ, διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο, ότι όλοι, και το είδατε και σήμερα, έτσι, μέσα από τις παρεμβάσει, όλοι διατηρούν τις ίδιες απόψεις. Υπερασπίζουν τι αρχές τους, υπερασπίζουν τα συμφέροντά του. Μα με αυτόν τον τρόπο δεν θα σημειώσουμε πρόοδο. Γιατί, γιατί Εάν μετά από την ανάλυση, αν, η ανάλυση είναι ίδια, η διάγνωση είναι ίδια και το 92 και το 98 και το 2002. Σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα προβλήματα είναι ε, ε, πολύ περισσότερα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Σήμερα η ευρωπαϊκή αγορά σε ποσοστό 62% εφοδιάζεται από τις εισαγωγές. Στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 μόλις το 20% προέρχονταν τις εισαγωγές. Χάνουμε την αγορά. Σήμερα ε, τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ε, πρέπει να σας πω ότι ε, ε, ε, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνονται νέα πλοία, ούτε σε επίπεδο βιοτεχνικό, γιατί ε, δεν είναι αποδοτική αλία. Τα προβλήματα λοιπόν είναι πολύ πιο σοβαρά σήμερα. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξουν πλέον μερικές λύσεις. Δεν μπορεί να υπάρξουν λύσεις που απλά και μόνο να απαλύνουν τα προβλήματα. Πρέπει να είναι φιλόδοξες οι λύσεις, πρέπει να είναι επί της ουσίας. Αυτή, ο απολογισμός, αυτή η διάγνωση ε, είναι κάτι που μα οδηγεί στο συμπέρασμα. Επίγει να λυθούν τα προβλήματα γιατί έχουμε την κρίση. Την κρίση θα τη βρούμε μπροστά μα και απαιτούνται επίγοντα μέτρα και επίγουσε λύσει. Τελευταία παρατήρηση. Η ανάλυση που κάναμε με βάση τη διάγνωση τη κατάσταση μα οδηγεί και σε ένα άλλο συμπέρασμα, το οποίο είναι θεμελιώδε. Δεν πρόκειται να βρούμε λύσει απομονωμένε. Δηλαδή, τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα οι απορρίψει, ε, η σχετική σταθερότητα, η μέθοδο διαχείριση, ε, η αποκέντρωση στι αποφάσει, ε, τα ITQ, όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν μεμονωμένα και να αποτελέσουν αντικείμενο μεμονωμένη διαπραγμάτευσης. Μα αν δεν λύσουμε το πρόβλημα τη υπεραλίευση, πώ θα συμφωνήσουμε με τα ITQ. Δεν μπορεί να έχουμε αποκέντρωση τη διαχείριση αν δεν έχουμε πολιτική ελέγχου με κοινού στόχου και κοινή πολιτική. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική της σχετικής σταθερότητας αν η προβληματική εξακολουθεί ε, να ε, αναφέρεται ε, σε ψευδείς δηλώσεις και σε έλλειψη ελέγχου. Ορισμένοι ομιλητές μίλησαν για το γεγονός ότι σε ορισμένα είδη δεν, έχουν, δεν ελιεύονται 30%. Μα ναι, ναι. α, α, αφού, αφού δηλώνονται ψευδή στοιχεία... 38% δεν δηλώνονται σωστά από τα κράτη-μέλη. Άρα μη μιλάμε ε, μεμονωμένα για τα προβλήματα. Να βρούμε λύσεις συνολικές. Λύσεις που ε, να είναι σφαιρικές και φιλόδοξες. Τελευταίο μήνυμα. Η συζήτηση είναι, είναι, θα είναι μακρά και ελπίζουμε να φύγουμε από αυτή την ε, αυτιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι θεσμοί, τα κράτη-μέλη. Γιατί η μοναδική λύση είναι να δράσουμε γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα έχουμε τέταρτη ευκαιρία. Το έλεγα και τι προάλλε σε μια συνεδρίαση που είχαμε του εκπροσώπου του κλάδου. Εάν επιβεβαιωθεί η κρίση και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται και οι σημερινέ προοπτικέ επιβεβαιωθούν, ίσω δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να συζητήσουμε. Γιατί θα περιθωριοποιηθεί τόσο ο κλάδο που σας, είπα, κλείνουν διαρκώς επιχειρήσεις, δεν, γίνονται, ε, δεν ανοίγουν νέες, τα πράγματα επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα. Πρόεδρε, θα υπάρξει η πράσινη βίβλος μέσα σε λίγες εβδομάδες, πράσινο βιβλίο ε, κλασικό, σύμφωνα με την παράδοση, 30 σελίδες, σύντομο έγγραφο, όπου θα υπάρξουν θα, θα τίθενται ε, ερωτήσεις για προβληματισμό. Δεν θα υπάρξει διάγνωση. Δεν θα τοποθετείται η Επιτροπή. Θα ε, αναφερθούν ερωτήματα για προβληματισμό. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Εκεί θα έχουμε ευρεία διάγνωση πάνω ε, από 500 σελίδες ε, που θα συμπεριλάβουμε και 30 κλαδικές μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Έτσι ώστε όλοι σας, ο κλάδος, όλοι οι εμπλεκόμενοι, ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην πολιτική να έχουν κοινή πληροφόρηση, άλλες φορές κριτική, άλλες φορές ανοίγοντας δυνατότητες. Πάντως όλα αυτά αυτό, ε, ε, αυτή, αυτός ο, ο ανοιχτός προβληματισμός θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους, να τους θέσουμε τους στόχους και να τους πετύχουμε. Δεν θα πρέπει να, ο καθένας να ε, περιχαρακώνεται στις θέσεις τους, γιατί σε αυτή την περίπτωση, όπως σας είπα, ίσως είναι η τελευταία φορά που συζητάμε το όλο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους σας, γιατί με βοηθήσατε ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να τελειώσουμε έγκαιρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους διερμηνείς, λέει Πρόεδρος, για την εργασία τους όλη αυτή ε, την ακρόαση και που μας έδωσαν και πέντε λεπτά χάριτος. Ε, σας ευχαριστούμε όλους. Ραντεβού λοιπόν με τα μέλη της Επιτροπής για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας αύριο από τις 9 το πρωί που θα έχουμε τη συνεδρία του Ινιστών. Σας ευχαριστώ.